Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε αυτή τη σημαντικότατη απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε, για την οποία έχουμε στη διάθεσή μας 3,5 ώρες. 3,5 ώρες εργασιών. Θα είμαστε εδώ στις 18.30. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι η ακρόαση διαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Ανοιχτό διαδίκτυο, ενιαία ευρωπαϊκή αδειοδότηση, φάσμα και περιαγωγή. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, ώστε να ανακτήσουμε και τα ελάχιστα λεπτά που χρειαστήκαμε για να καθίσουμε όλοι και θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Πιλάρ Καστίγιο. Είναι η συγγήτριά μα για τα θέματα τηλεπικοινωνιών, για το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Παρακαλώ, Πιλάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε όλοι σα και από μένα σε αυτή την ακρόαση που αφορά την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά για τις τηλεπικοινωνίες. Συμπεριλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, όπως είπε και η πρόεδρος μας. Θα τα δούμε ένα κεφάλαιο, λοιπόν, σε στήλες. Το πρώτο αφορά το ελεύθερο διαδίκτυο και χωρίς περαιτέρω σχόλια να ξεκινήσουμε πιστεύω με, τέσσερις, με τρεις ομιλητές. Πρώτος είναι ο Ερικ Ντεβρόκ, έχουμε και τον Μπενουά Λουτρέλ, Γενικό Διευθυντή της ΑΡΣΕΠ και μετά τον Γιάνν Βίσνερ, Υποδιευθυντή του ε, Γραφείου Συνδέσμου ARD. Παλακαρό, κύριε Ντεβρούκ, ξεκινήστε εσείς. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Σαρτόρη και την εισηγήτρια κυρία Τερκαστήγιο, που διοργάνωσαν αυτήν την δημόσια ακρόαση σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντες από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Θα μιλήσω σήμερα για την ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ, το διαδίκτυο και τις σχετικές διατάξεις της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να λειτουργεί το μηχάνημα των διαφανειών. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η εμπειρογνωμοσύνη των προμηθευτών διαδικτύου είναι απαραίτητε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκε των πελατών μα. Ασχολούμαστε με τη σταθερή και κινητή παροχή υπηρεσιών ε, πρόσβαση στο διαδίκτυο με τι υπηρεσίε ADSL, 3G και το Medium. Έχει πολλαπλασιαστεί η ταχύτητα πρόσβασης ε, στο διαδίκτυο και το αποτέλεσμα είναι ότι βιομηχανία μας, ε, η εταιρεία μας μάλλον, επενδύει το 10% του κύκλου εργασιών της ετησίως στα θέματα αυτά. Δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε τις, να κατασκευάζουμε τις υποδομές και είμαστε από τις εταιρείε με τις καλύτερες, με τις περισσότερο, με τις υψηλότερες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών μας. Τώρα, υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες που προτείνεται. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο που επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη να φτάσει σε ένα τελείωτο πλούτο διαδικτυακών υπηρεσιών αλλά και η διαχείριση των υπηρεσιών ε, στην ε, καθημερινή κυκλοφορία στο διαδίκτυο ώστε να γίνεται βέλτιστη δυνατική χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνει το διαδίκτυο. Αυτό ονομάζεται Best Effort Routine, η ρουτίνα των ε, βέλτιστων προσπαθειών. Έπειτα, πέρα από την πρόσβαση, οι προμεθευτές του διαδικτύου προτείνουν και ειδικέ υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο επίπεδο ε, υπηρεσιών, όπως η τηλεφωνία ή οι υπηρεσίες ε, τηλεόρασης, IP, όπως έχουν ονομαστεί. Αυτό είναι ωφέλιμο για τους τελικούς χρήστες, γιατί γίνονται οικονομίες που ωφελούν και τις δύο πλευρές, δηλαδή επενδύσεις σε μονάδες για την βελτίωση της ποιότητας της τηλεοπτικής ε, παροχής, βελτιώνει και την ταχύτητα του διαδικτύου, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών υποδομών. Σε έναν κόσμο ανταγωνισμού, οι τηλεπικοινωνίε και οι εταιρείε τηλεπικοινωνία που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν προκειμένου να είναι ελκυστικέ για του πελάτε του, για του καταναλωτέ. Δεν έχουν όλοι οι πελάτε το ίδιο βαλάντιο, ούτε χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε με τον ίδιο τρόπο και ταυτόχρονα. Επίση, δεν έχουν ε, την ικανότητα να έχουν πρόσβαση στι ίδιε υπηρεσίε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει με τις ίδιες υποδομές μια ποικιλία υπηρεσιών που να παρέχεται. Η διαχείριση της κυκλοφορίας είναι επίσης κρίσιμη σημασία για να υπάρχουν καλές ποιότητας υπηρεσίες σε λογικές τιμές. Οι Orange σε γενικέ γραμμέ ε, είναι υπέρ των διατάξεων ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ, ε, στο διαδίκτυο, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά με τέσσερι διευκρινήσει. Οι πελάτε, οι καταναλωτέ χρειάζονται σαφεί, δίκαιε και αξιόπιστες πληροφορίες για την πρόσβαση χωρίς να υπερφορτώνονται με περιτές ε, πληροφορίες. Οι τροπολογίες που προτείνονται από ε, τον κύριο Χάρμπορ για την ταχύτητα πρόσβαση στο διαδίκτυο ε, ευθυγραμμίζονται περισσότερο με την πραγματικότητα που ισχύει στον κόσμο του ίντερνετ. Δεύτερη διευκρίνηση. Η προτινόμενη αρχή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας είναι λογική. Από την άλλη όμως λιγότερο αποδεκτές πρακτικές δεν θα πρέπει να εξαλειφθούν, θα πρέπει να υπάρξει η πρόληψη για την ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση στο διαδίκτυο και όχι απλώς να φροντίσουμε να την εξαλείψουμε. Η δυναμική ανακατανομή η σωστή μάλλον κατανομή είναι σημαντική για την ε, καλύτερη διαχείριση του κόστους και των ε, προσπαθειών που γίνονται. Και θα πρέπει να επιμείνουμε σε έναν ορισμό των ειδικών υπηρεσιών. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο κύριος Χάρμπορ με τη διατύπωση που προτείνει αποσαφηνίζει ότι οι ειδικές υπηρεσίες παρέχονται από τους φορείς τηλεπικοινωνιών βάσει των ελέγχων πρόσβασης στην αγορά ώστε να είναι σαφής η ποιότητα που προσφέρεται στους πελάτες μέσω της εμπειρίας που διατίθεται. Ε, τέλος, στηρίζουμε την έκθεση της δικής σας συγγήτριας που προτείνει ένα κατάλογο με προτεραιότητες για την επόμενη αναθεώρηση του σχετικού πλαισίου και περιμένουμε η διαδικασία να ε, εκκινηθεί πριν από τα τέλη του 2014. Όταν αρχίσει αυτή η μελλοντική αναθεώρηση θα πρέπει να δούμε αν θα ισχύει η αρχή ίδια πρόσβαση ίδιες υπηρεσίες. Γιατί εντωμεταξύ οι ειδικέ υπηρεσίε θα πρέπει να είναι αλληλοσυμπληρωματικέ, ώστε οι υπηρεσίε διαδικτύου να μπορούν να, να αξιοποιηθούν από τους φορείς τηλεπικοινωνιών που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την ηλεκτρονικό ιδιωτικό βίο ή κανόνες για τις κατεπήγουσες καταστάσεις ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές αλλά και να υπάρχει διακυβερνητική ασφάλεια για θέματα προσωπικού και ιδιωτικού βίου. Επίση, να αποφύγουμε τον αθέμετο ανταγωνισμό ή την στρέβλωση τη αγορά. Μια λύση θα είναι να εξυγχρονίσουμε τον ορισμό των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το πλαίσιο του 2002 που έχει γίνει απορχαιωμένος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την πολύ αστιασμένη παρουσίασή σας και δίνω τώρα το λόγο τον κύριο Μπενουά Λουτρέλ Γενικό Διευθυντή της ΑΡΣΕΠΑ από τη Γαλλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ε, δεν μιλάω εξ ονόματος της ΑΡΣΕΠΑ, αλλά του ΡΕΣΕ, δηλαδή ε, εξ ονόματος του Οργάνου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο έτσι ώστε να μιλήσω για την ουδετερότητα των δικτύων να θυμίσω την τοποθέτηση της ΟΡΕΣ όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων, πράγμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό. Και μετά θα σας πω ποια είναι η ανάλυση μας όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αρχία αρχή αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι θεμελιώδες δικαίωμα ε, των πολιτών της Ευρώπης από το τέλος του προηγούμενου αρχή του Τωρινού ε, και ε, η δημόσια θέση που λέει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό το κεκτημένο είναι ουσιώδου σημασία. Πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι operators των τηλεπικοινωνιών είναι μέρος της λύσης. Σήμερα ε, έχουμε μεγάλη επιτυχία στο ίντερνετ και την χρήση του ίντερνετ και αυτό ε, διότι η βιομηχανία της τηλεπικοινωνίας ε, κατάφερε να απαντήσει σε, αυτό το αίτημα και επομένως προώθησε την διαδικασία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βεβαίως ε, δεν ε, υπάρχει παρθενογέννηση όσον αφορά τις ρυθμιστικές αρχές ε, και επομένως υπάρχει μία νόμιμη ανησυχία σχετικά με την διαχείριση του δικτύου και κατά πόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο ανοιχτό ίντερνετ. Το είπαμε και αυτό επανειλημμένα ότι η διαχείριση της κυκλοφορίας στα δίκτυα είναι εγγενώς συνδεδεμένη με τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υπηρεσίες των ε, παρόχων τηλεπικοινωνικών ε, υπηρεσιών και βεβαίως ε, που δεν παράγουν μόνο την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό προϋποθέτει ότι είναι νομιμοποιημένη η διαχείριση της κυκλοφορίας στο δίκτυο. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες πρακτικές οι οποίες μπορεί να είναι προβληματικές και κατά αυτή την άποψη βεβαίως μπορεί να χρειάζεται κάποια δημόσια δράση. Στα παρόντα πλαίσια εμείς σαν οργανισμός, σαν υπηρεσία έχουμε προετοιμάσει μια θέση με σημεία δράσης. Πρώτον να αφήσουμε την λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς. Ξέρουμε ότι η αγορά λειτουργεί καλά σε αυτές τις περιπτώσεις και επομένως στο ΟΡΕΣ θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει πραγματική ουσιαστική διαφάνεια, να Ξέρουμε δηλαδή ποια είναι ε, η προσφορά των ε, διαφόρων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ε, στον πολίτη έτσι ώστε αυτός να μπορεί να επιλέξει και ενδεχομένως να αλλάξει και πάροχο. Αυτό βεβαίως σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα πρέπει ο πελάτης να μπορεί να αλλάξει πάροχο χωρίς ψηλό κόστος. Δεύτερο σημείο, επιτήρηση από πλευράς των ρυθμιστών έτσι ώστε να να μελετηθούν ε, οι διάφορες πρακτικές των ε, ε, παρόχων Telecom. Ε, και βεβαίως το τελευταίο σημείο ήταν να πούμε ότι όντω ο ρυθμιστής πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει, αλλά ε, κάνοντας ανάλυση αναπερίπτωση έτσι ώστε να είναι πραγματική ε, η ανάλυση της πρακτικής και το κατά πόσον αυτή η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί ή όχι πρόβλημα. Να υπάρχουν σκοπιμότητες, σκοπιμότητες που οδηγούν σε πρακτικές οι οποίες είναι σωστές, άλλες λιγότερο σωστές, μπορεί να υπάρχει καταχρηστική διακριτική μεταχείριση ε, ε, ε, συγκεκριμένες δοκιμές λοιπόν γίνονται έτσι ώστε να παρέμβει ο ρυθμιστής όταν και εφόσον είναι απαραίτητο. Σε γενικές γραμμές η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει οικοδομηθεί πάνω στην ίδια αντίληψη και την ίδια βάση. Είναι γεγονός ότι εμείς σαν υπηρεσία δεν δείξαμε τρομερό ενθουσιασμό στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξ αρχής, αλλά στην προκείμενη περίπτωση περίπτωση πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Βεβαίως, όπως και σε όλα τα κείμενα που μπορεί να ε, υποβάλει ένας συνομοθέτης, Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωση, αλλά σε γενικέ γραμμέ είμαστε ικανοποιημένοι. Οι εξειδικευμένε υπηρεσίε, οι υπηρεσίε πρόσβαση στο ίντερνετ ε, ξεκαθαρίζονται, διευκρινίζονται ε, σαφώ. Η ύπαρξη ειδικών εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν δυναμητίζει τις αρχές πρόσβασης στο ίντερνετ που πρέπει να είναι απολύτως ανοιχτές. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας, δυνατότητας αλλαγής παρόχου κτλ. Βλέπουμε όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για μια καλή πρόταση. Για να ολοκληρώσω ε, σύντομα θα κάνω ε, κάποια σχόλια. Πρώτον, το νομικό εργαλείο οδηγία ή κανονισμός. Εδώ προτείνεται κανονισμός. Ε, θεωρούμε ότι ε, μπορεί να είναι το προσήκον εργαλείο εάν και εφόσον ο κύριε κεντρικός στόχος ε, της δημόσιας πολιτικής, συγγνώμη, της υπηρεσίας δημόσιας ωφέλειας εάν αναγνωριστεί. Θα πρέπει να υπάρχει άλλωστε και η απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής στις διάφορες καταστάσεις. Η Ευρώπη είναι αυτή που είναι ε, υπάρχει επίσης και μία αρμονική κατά την άποψή μας ρύθμιση των αγορών τηλεπικοινωνιών ε, αλλά ε, χρειάζεται εξατομίκευση κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία η οποία θα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεμονωμένες πρακτικές και στις εξειδικευμένες καταστάσεις. Ε, θα πρέπει να δούμε πρακτικές οι οποίες ε, δεν πρέπει να είναι καταχρηστικές, οι οποίες στο παρελθόν ενδεχομένως δεν ήταν και ίσως έχουν γίνει τώρα λόγω της παρουσίας του ε, διαδικτύου και επομένως πρέπει να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα προσαρμογής και στις ενδεχόμενες αλλαγές οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω σχετικά με την ε, ε, αλληλόδραση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες ε, υπηρεσίες καθώς επίσης και μεταξύ Μπερέκ και ρυθμιστών. Είμαστε πεπισμένοι ότι από αυτού η Κομισιόν ε, είναι, ε, έχει σωστά αντιμετωπίσει το θέμα ε, και αυτό διότι βασίστηκε σε την τεχνογνωσία της δικής μας υπηρεσίας και κατάλαβε τα σημεία επί των οποίων πρέπει να υπάρχει ευελιξία και τα σημεία επί των οποίων δεν χρειάζεται τόση πολύ ευελιξία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε όλες τις πρακτικές Τώρα το κατά πόσον επειδή το ωραίο συμφωνεί με τι πρακτικέ αυτές, αυτές είναι σωστέ ή όχι, το αφήνω στη δικιά σας ε, ε, κατανόηση. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, ο επόμενο συμμετέχων στο πάνελ, ο κύριος Βίσνερ, υποδιευθυντής του Γραφείου Συνδέσμου ARD. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σήμερα στην ακρόαση που διεξάγεται για να μπορέσουμε να σας εξηγήσουμε την χρήση του ARD. Το διαδίκτυο και για μας γίνεται όλο και πιο σημαντικός τρόπος ε, ε, μετάδοσης του περιεχομένου μας και για να ασκήσουμε τα καθήκοντα που μας αναθέτει ο Εθνικός Νομοθέτης και για να φτάσουμε μέχρι το κοινό μας. Έχουμε το ανοιχτό διαδίκτυο που παίζει σημαντικό ρόλο στην ελευθερία έκφρασης, ελευθερία ενημέρωσης, στην γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία και στην πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας. Σε πιο γενικό επίπεδο ως πάροχοι περιεχομένου, συμφωνούμε με άλλους παρόχους περιεχομένου, σε ό,τι αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα του ίντερνετ. Η ουδετερότητα του δικτύου είναι προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί έντιμος και ζωντανός ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων περιεχομένου, καθώς και για την είσοδο νέων παικτών. Ο ανοιχτός χαρακτήρας και η μη διακρίσεις στο διαδίκτυο είναι βασική μοχλή για ανανέωση και για οικονομική αποδοτικότητα καθώς και για την διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων. Από την σκοπιά μας είναι λοιπόν ουσιώδες να πούμε ότι το ανοιχτό ίντερνετ πρέπει να είναι ο κανόνας και ότι οι δικευμένες υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελέσουν την εξαίρεση και να μην παρεμβαίνουν στο ανοιχτό ίντερνετ. Δεν είμαστε καταρχήν κατά των ε, εξειδικευμένων υπηρεσιών, παρόλο που κάποιοι ορισμοί στην πρόταση για μας δεν είναι απόλυτα σαφείς, διότι και εμείς χρησιμοποιούμε διαχειριζόμενες υπηρεσίες, managed services, άλλωστε εντάσσεται και ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να φτάσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο και με τις ε, πλατφόρμες τηλεόρασης κλπ. Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι πολίτες πρέπει πάντοτε να διαθέτουν την δυνατότητα άνευ περιορισμών πρόσβασης σε όλα τα περιεχόμενα του ανοιχτού δικτύου. Αυτή πρέπει να είναι η βάση. Αυτό ιδίως έχει σημασία σε ένα κόσμο που οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών καθετοποιούνται όλο και περισσότερο, που υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος της υποδομής του διαδικτύου, όπου προσφέρονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες και μάλιστα και ορισμένες από αυτές διαθέτουν πλέον και αποκλειστικά δικαιώματα στο περιεχόμενο. Αυτό προκαλεί τον κίνδυνο οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών να προβούν σε διακρίσεις κατά περιεχόμενων άλλων παροχών οι οποίοι βασίζονται στην δική τους υποδομή για να ε, διαδώσουν το περιεχόμενό τους. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να συμβεί, είναι προφανές. Γι' αυτό εργαζόμαστε για να θεσπιστούν νομικές διατάξεις που θα προφυλάσσουν απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Θεωρούμε πάντως ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Πρώτα, ο ορισμός των υπηρεσιών πρόσβασης διαδικτύου δεν είναι, οι ορισμοί αυτοί δηλαδή δεν είναι αρκετά ξεκάθαροι. Νομίζουμε ότι οι ορισμοί που προτείνει η Μπερέκ είναι πιο σαφείς. Επιπροσθέτως, η αρχή της βέλτιστης προσπάθειας πρέπει να κατοχυρωθεί και πιστεύουμε ότι ο κύριος Χάρμπορ στην, στο σχέδιο πρότασής του κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερο, είναι κρίσιμη σημασία να υπάρξει διαφάνεια ανάμεσα στο ανοιχτό διαδίκτυο και στις λεγόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Το διαδίκτυο πρέπει να παραμείνει ο κανόνας. Δεν επιτρέπεται να γίνει εξαίρεση. Αν μου επιτρέπετε να δηλώσω το εξής, όλοι έχουμε αναγνώσει το κείμενο και βεβαίω η ανάγνωση του κειμένου φαίνεται να γίνεται διαφορετικά για τον καθένα τουλάχιστον κατά ορισμένα σημεία. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και σε αυτό το θέμα. Τρίτο, στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να δούμε κάποιες διευκρινήσεις για το άρθρο 19 για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Γιατί το άρθρο αυτό στοχεύει πιο μακροπρόθεσμα σε νέους τύπους online υπηρεσιών. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ άρθρου 19 και άρθρου 23 μαθαίνω ότι η συγκήτριά σας κινείται προς την κατεύθυνση αυτή με την διαγραφή ορισμένων παραπομπών του άρθρου 19. Τέταρτο, δοθέτων των κινδύνων της καθετοποίησης των operator, η αρχή της μη διακρίσεως πρέπει να ενισχυθεί. Τέλος, όταν παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των ειδικευμένων υπηρεσιών στο ανοιχτό ίντερνετ, όπως ορίζει το άρθρο 24 της προτάσεως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα αποτελέσματα των ειδικευμένων υπηρεσιών επί της πολιτιστικής ποικιλία, αλλά και επί της ελευθερίας εκφράσεως, ενημερώσεως και πολυφωνίας των μέσων. Διότι το διαδίκτυο δεν είναι κρίσιμο μοναχά για την οικονομία μας, σήμερα είναι ουσιώδες και για τις δημοκρατίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Ε, εγώ και άλλοι συνάδελφοι θα παρέμβω μετά. Η κυρία Τροτμάν όμως πρώτη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι για να βεβαιωθούμε ότι γίνονται σεβαστές οι απαιτήσεις περί διαφάνειας ε, δεν αρκεί να αλλάζουμε προμηθευτή. Γι' αυτό έγινε αναθεώρηση του πακέτου το 2009. Ήδη τότε υπήρχε συνένεση για να γίνουν οι σχετικέ αλλαγέ, αλλά τελικά αυτό δεν εξαρκούσε για να υπάρξει ουδετερότητα του διαδικτύου. Νομίζω λοιπόν ότι ένα μέρος της συζήτησης που έχουν στηρίξει με τις παρεμβάσεις τους και οι συμμετέχοντες τους οποίους ευχαριστώ έχει να κάνει με την κυκλοφορία στο διαδίκτυο και πώς ακριβώς την ορίζουμε πώς επιτρέπουμε να διαμορφωθεί. Εάν η διαχείριση της κυκλοφορίας, της κίνησης στο διαδίκτυο ε, έχει να κάνει και με θέματα συμφόρησης, δεν μας φαίνεται δυνατό να αφήσουμε τους προμηθευτές χωρίς ε, εγγυήσεις, χωρίς προστατευτικά δίκτυα. Θα πρέπει να γίνουν κάτι σαν ε, φύλακες Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πάμε ίσως λίγο πιο μακριά στην πρότασή μας. Μια δεύτερη πτυχή που θέλω να τονίσω έχει να κάνει για τις υπηρεσίες τις οποίες διαχειριζόμαστε. Δεν διαφωνώ επί της αρχής, είναι μια δυνατότητα που θα πρέπει να την διερευνήσουμε. Υπό την αίρεση όμως γεγονότος ότι το best effort θα διατηρηθεί. Εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε τη συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου και το best effort δεν θα πρέπει να να μπει στο παρασκήνιο, ε, να περάσει σε δεύτερη μοίρα μάλλον και να το διατηρήσουμε ως προτεραιότητα. Γιατί εάν με σαφείς ορισμούς ε, εγγυηθούμε αυτό το best effort και με έναν μηχανισμό που θα λειτουργεί σωστά, τότε μπορεί και να έχουμε αποτελεσματικότητα στις διατάξεις που προτείνονται. Ιδάλλως μάλλον όχι. Αυτά ήθελα να επισημάνω και εγώ στους παρεμένοντές μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Κατρίν. Άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Δεν βλέπω το όνομά σας. Ναι, έχω ερώτηση για το best effort και τη σχετική αρχή. Αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις προσπαθεί να κάνει κανείς ό,τι καλύτερο μπορεί για την αποστολή δεδομένων. Εάν όμως έχει κανείς μια δυνατότητα ε, να αν έχει ιδιαίτερες ε, δυνατότητες ως προς το φάσμα. Ε, υπάρχει πάντοτε αντίφαση μεταξύ των ειδικών υπηρεσιών και των υπολείπων. Οι ειδικέ υπηρεσίες μάλλον είναι πιο επικερδείς. Οπότε οποιοδήποτε προμηθευτής διαδικτύου ε, θα προτιμά τις ειδικές υπηρεσίες από το ελεύθερο διαδίκτυο. και η αρχή της ε, βέλτιστης προσπάθειας δεν θα εγγυάται κάποια συγκεκριμένη ποιότητα υπηρεσιών. Οπότε και εγώ ως οικονομολόγος θα περίμενα να υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα από την απελευθέρωση του διαδικτύου εν τέλει. Τι άποψη έχετε εσείς, πώς μπορεί να ε, επιληθεί αυτή η σύγκρουση συμφερόντων. Ε, yes, um, I'm sorry because Δεν σας ανεγνώρισα αμέσως και δεν είπατε το όνομά, το όνομά σας. Είστε οι εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών. Δεν είστε γενικό κοινό δηλαδή, είστε Επιτροπή Περιφερειών και επίσης ο συνάδελφός μας απέναντι. Ερώτηση. Ο κανονισμός λέει ότι η πάροχη Telecom δεν κάνουν διακριτική μεταχείριση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, οφείλει να εξασφαλίζεται η ουδετερότητα του δικτύου. Η ερώτησή μου προς τους provider είναι οι ειδικευμένες υπηρεσίες μου φαίνεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν μόνο όταν προσφέρεται τις ειδικευμένες υπηρεσίες με καλύτερη ποιότητα κλπ. χωρίς να προβείτε σε αρνητική διάκριση για την χρήση του διαδικτύου. Είναι δυνατόν αυτό ή είναι εσφαλμένη αυτή η νοοτροπία. Θα μιλήσω ισπανικά τώρα. Νομίζω ότι θα μπορέσω να μιλήσω και συντομότερα τότε. Έχω λοιπόν από το εξή. Αφού πρώτα ευχαριστήσω και τους ε, αγορητές μας, πρόκειται για ένα μέρος της προτάσεως της Κομισιόν που έχει ξεκινήσει, θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι το τμήμα εκείνο της προτάσεως της Κομισιόν που συγκέντρωσε και την μεγαλύτερη υποστήριξη από τους διάφορους τομείς που συνδέονται με τη βιομηχανία ICT και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στο διαδίκτυο. Όπως μας εξήγησε ο εκπρόσωπος του γαλλικού ρυθμιστή, της Γαλλικής Ρυθμιστικής Αρχής υπάρχει συμφωνία και υποστήριξη από την ΠΕΡΕΚ και η Κομισιόν συμφωνεί. Και είναι σημαντικό να το αντιληφθούμε αυτό. Διεξήχθη ανάλυση στη βάση των πληροφοριών που ήταν διαθέσιμες και μια, κοινή, μια μεικτή επιτροπή μάλλον κατέληξε σε συμπεράσματα όπως είπε και η ρυθμιστική αρχή, τα συμπεράσματα αυτά απηχούνται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι σημαντικό. Εξετάζουμε τα θέματα από σκοπιά επιχειρηματική αλλά και νομοθετική. Εξετάζουμε την νομοθεσία του ευρωπαϊκού επίπεδου όπως αυτή εφαρμόζεται από τους εθνικούς ρυθμιστές. Δεν είναι ασήμαντο λοιπόν το θέμα όταν προβαίνουμε εμείς στη δική μας αξιολόγηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι τότε θα λάβουμε υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις. Θεωρούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι στέρεα. Χρειαζόμαστε διευκρίνηση σε ορισμένα θέματα για να διασφαλίσουμε ότι πρόσβαση στο διαδίκτυο θα διαθέτουν όλοι. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο ανοιχτό και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και στα άτομα και στις επιχειρήσεις και στους πολιτές και στους αγοραστές και στις επιχειρήσεις και στους προμηθευτές. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε, να αφαιρέσουμε κάθε είδους διάκριση μέσα από το διαδίκτυο. Είναι αληθές επίσης ότι ίσως ένα αριθμό επιχειρήσεων τελικά να μην έχει τον ίδιο βαθμό πρόσβασης. Εάν όμως προβούμε σε υπερβολική ρύθμιση νομίζω θα αναχαιτήσουμε την πρόοδο και στο παρόν αλλά και κυρίως στο μέλλον. Συνεπώς θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ισορροπία σε κάθε μορφή ρύθμισης. Εν προκειμένου δε καταστρώνουμε ένα κατάλογο αρχών που να διέπουν τους κινδύνους του διαδικτύου. Αυτό βρίσκω ότι είναι σημαντικό. Προσωπικά, στην έκθεσή μου έχω υποστηρίξει τις προτάσεις της Κομισιόν και προσπαθώ να τονίσω και να τονώσω την αρχή της, των μη διακρίσεων. Και προτείνω μέτρα για να ενισχυθεί η αρχή παράληψης διακρίσεων. Εάν σημειωθεί διάκριση, τότε πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω την αρχή της βέλτιστης προσπάθειας. Είναι δύσκολο όμως να προχωρήσουμε πέρα από κάποιες αρχές. Όπου υπάρχει διάκριση, το θέμα θα πρέπει να παραπέμπεται ιδίως στους εθνικούς ρυθμιστές, να εφαρμόζουν τους μηχανισμούς που προβλέπονται επιτόπου στις χώρες μέλη. και να εξαντλούνται τα, η διοικητική και δικαστική διάβλη σε αυτό το επίπεδο πρώτα. Θα έχουμε μπροστά μας το ανοιχτό διαδίκτυο που θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες πρόσβαση σε όλους. Αλλιώς πρόκειται για αποτυχία. Έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να αποτελματοθούμε μέσα στα ατελείωτα εάν και ναι μεν αλλά κτλ. Χρειαζόμαστε κάποια μορφή ρύθμισης, χρειάζεται να τονίσουμε την αρχή της εξάλληψης πάσης διακρίσεως και αυτή τελικά είναι η προσωπική μου γνώμη. Βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα πράγματα αυτά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Ήτρε και τελικά παραμένω αισιόδοξη ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε συμφωνία όπως έπραξε η Μπερεκ και η Κομισιόν. Θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ε, με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν. Γνωρίζω ότι υπάρχουν τώρα ορισμένε ερωτήσεις προς τους προσκεκλημένους ομιλητές και θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Ποιοςδήποτε εξημών επιθυμεί να απαντήσει η κυρία Τρότμαν, έθεσε μια ερώτηση, ο κύριος Κρόιτσμαν επίσης, καθώς και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, κάποιες ερωτήσεις αφορούσαν την αρχή της βέλτιστης προσπάθειας, του best effort. Νομίζω ότι όντως όλος ο κλάδος έχει βασιστεί σε αυτή την αρχή και όλες οι προσφορές σε αυτήν ε, έχουν ε, σχεδιαστεί, βάσει αυτής έχουν σχεδιαστεί. Έτσι έχει σχεδιαστεί και όλη μας η οικονομική διοργάνωση. Πρόκειται για ένα σύστημα που ούτως ή δεν είναι ανεξέλεγκτο. Λειτουργεί μάλιστα εύρυθμα, διότι ανταποκρίνονται σωστά και αγορές και θα πρέπει ο ο τελικός χρήστης, να γνωρίζει ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Έτσι, το σχέδιο του κανονισμού, όπως έχει υποβληθεί, ενισχύει αυτήν την ε, εναλλακτική με την πρόταση για δείκτες ποιότητας. Επίση, εφόσον διαπιστωθούν αρνητικέ τάσει στι αγορέ ή καταστροφικέ έστω προ την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να καταρρεύσουν, τότε ο ρυθμιστή μπορεί να παρέμβει, επιβάλλοντα μια ελάχιστη ποιότητα για τι υπηρεσίε. Αλλά παραμένει τρίτο το γεγονό ότι ω τώρα η ιστορία διαρκώ μα αποδεικνύει ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ολοένα και πιο ε, έντονη. Βλέπουμε ότι σε αυτό επενδύουν οι προμηθευτέ και ότι υπάρχει σοβαρή ζήτηση, μεγάλη ζήτηση. Όσο μεγαλύτερη ζήτηση υπάρχει, τόσο περισσότερη ταχύτητα απαιτείται επίση. Και μέχρι τώρα είναι θετική αυτή η αναλογία και η σχέση με μηχανισμού που ενισχύονται και θα ενισχυθούν περαιτέρω από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ούτω ή άλλω σημαντικό είναι να την ε, αντιληφθούμε αυτή την ε, ε, έννοια της βέλτιστης προσπάθειας, γιατί αυτή καθορίζει την οικονομική αξία της προσφοράς. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν με μια προσφορά μηδενική σε αυτή την περίπτωση. Εδώ μιλάμε για 30 ευρώ σε μια βασική παροχή, τη βασική υπηρεσία που προτείνεται. Αλλά το δικαίωμα του Ευρωπαίου ε, καταναλωτή να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο θα απειλεί το, εάν γινόταν κάτι τέτοιο. Κατάρρευση των τιμών και της ποιότητας. Τώρα δεύτερο ερώτημα για την διαχείριση της κυκλοφορίας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη έλλειψη προστατευτικών δικτύων λόγου χάρη, αλλά ούτε και περιορισμούς. Θα πρέπει να μην είμαστε υπερβολικοί στη ρύθμιση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυναμικές τάσεις αυτή τη στιγμή και όσο περισσότερες όσο περισσότεροι φραγμοί εξαλείφονται εξαλείφονται φυσικό το τρόπο, τόσο περισσότερο αναπτύσσονται τα δίκτυα και γίνονται πιο σύγχρονα, όπως το 4G στη Γαλλία που έχει λάβει ήδη μεγάλες διαστάσεις. Η δυνατότητα λοιπόν του καταναλωτή να επηρεάσει αυτό στις αγορές είναι πολύ μεγάλη. Όταν οι αγορές αναπτύσσονται, οι πελάτες αλλάζουν και επίπεδο υπηρεσιών. Και εμ, κάπως έτσι δημορφώνεται αυτή η σχέση. Είναι ένα αστιακό σημείο αυτό. Επίσης, η νομοθεσία, όπως προτείνεται, προτείνει μια συγκεκριμένη αρχή, λέγοντας ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να παραμένει ελεύθερη, αλλά το κόστος της διαχείρισης των υπηρεσιών είναι μεγάλο. Υπάρχει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε έτσι θα πρέπει να δοθούν και μια σειρά από διαβαθμισμένες ε, απαντήσει αυτές τις ανάγκες για να υπάρχουν και απαραίτητες νομικές ε, εγγύησεις και διαδικασίες. Τώρα, για το αν θα υπάρχει διαχείριση των ε, υπηρεσιών ή ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όχι, δεν είναι το ένα ή το άλλο. Η πρώτη ειδική υπηρεσία είναι το τηλέφωνο, ούτως ή άλλως. Κανείς δεν φαντάζεται όταν αγοράζει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ε, ελεύθερο, δεν μπορεί να φανταστεί ότι η πρόσβαση στο τηλέφωνο θα είναι περιορισμένη. Όλοι θέλουν όταν κάποιος μπορεί να δει τον Μπόργεν στην τηλεόραση στο σπίτι, να μπορεί ταυτόχρονα κάποιος άλλος με στο ίδιο σπίτι να κάνει και ένα κατεπήγον τηλεφώνημα. Ε, οι ειδικέ λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες και η εξέλιξή τους μας δείχνουν ότι πρέπει να τις προσφέρουμε. Δεν είναι καθόλου αθέμητες ε, από τις αρχές. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω στα γαλλικά. Και εγώ. Θα ήθελα και εγώ να δώσω ορισμένα στοιχεία απάντησης. Πρώτον, το ερώτημα το οποίο θέσατε σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις υπηρεσίες best effort. Αυτό νομίζω ότι είναι παραγωγικό με την έννοια ότι θα ήταν οικονομικό λάθος. Παίρνω ένα απλό παράδειγμα μεταξύ του IPTV ε, σε μια προσφορά triple play ε, και την υπηρεσία πρόσβαση στο ίντερνετ. Όταν δεν βλέπουν πολύ τηλεόραση ε, στο, στο σπίτι που έχει γίνει αυτή η σύνδεση. Η ικανότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ίντερνετ. Όταν λειτουργεί η IPTV, αυτή η τηλεόραση, ε, τότε η ικανότητα της, ε, του, του ίντερνετ ε, μειώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. εάν δεν χρειάζεται κοινή προσφορά, τότε κάνουμε μία προσφορά χωρίς τη τηλεόραση, αν δεν είναι αρκετή η δύναμη. Εάν θέλουμε συστηματικά να εξασφαλίζουμε το σύνολο της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 Ε, Όταν θέλουμε το σύνολο του φάσματος ε, για το ίντερνετ, τότε αφήνουμε την τηλεόραση. Ε, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα οικονομικό και ένα πρόβλημα επομένως αποδοτικότητας. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να είστε πολύ προσεκτικοί φαντάζομαι στις αποφάσεις που θα πάρετε όσον αφορά την ορολογία γιατί διαφορετικά βάσει αυτής της αντίληψης του best effort μπορεί τελικά να δημιουργήσει δημιουργηθεί οικονομικό πρόβλημα προζημίαν και των παρόχων αλλά τελικά και των καταναλωτών. Το δεύτερο σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι η ε, δυναμική διαχείριση καθώς επίσης και η ανάγκη αποφυγής, πρόληψης μάλλον, ε, των, ε, της συμφόρησης υπάρχουν δυνατότητες διαχείρισης κυκλοφορίας που θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στο τελικό κείμενο κατά την άποψή μας ε, και ε, προβλέπονται ε, όχι μονάχα η διαχείριση της κυκλοφορίας εφόσον προκύψει συμφόρηση αλλά η πρόληψη της συμφόρησης μέτρα δηλαδή τα οποία θα αποτρέψουν την συμφόρηση και επομένως θα επιτρέψουν μια πιο αποτελεσματική διαχείριση και επομένως θα ανταποκριθούν αποτελεσματικό γενικότερα στα αιτήματα των ε, ε, πελατών. Ε, και βεβαίως τελειώνοντας να πω ότι εμείς ως πάροχοι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μας απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα του ανοιχτού ίντερνετ γιατί πρόκειται βεβαίως για μια υπηρεσία η οποία ιδιαίτερως ενδιαφέρει όλους τους πελάτες. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γερμανικά μια σειρά από Το πρώτο που έθιξε η κυρία Τροτμάν για την διαφάνεια βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι και επαρκές. Σίγουρα οι ρυθμιστικές αρχές έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν εν προκειμένου, διότι μπορούν να κάνουν και συγκρίσεις των διαφόρων παρεχομένων υπηρεσιών. Όμως για τον μεμονωμένο καταναλωτή είναι δύσκολο να αντιληφθεί πού εντοπίζεται το πρόβλημα όταν βλέπει ότι έχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα προέρχεται από τον πάροχο περιεχομένου, από, τον, ε, από αυτόν που ε, διαχειρίζεται το, το διαδίκτυο, από το network capacity, από το router capacity. Ακόμη και αν κατανοεί πώς λειτουργεί κάποιος, παρόλα αυτά για τον μεμονωμένο καταναλωτή είναι πολύ δύσκολο να τα διακρίνει. Η διαφάνεια λοιπόν γνωρίζει όρια. Σίγουρα δεν είναι η λύση του προβλήματος. Δεύτερο που έθιξε πάλι η κυρία Τρότμαν η σχέση των διαχειριτών, των ε, ε, διαχειριζόμενων υπηρεσιών με το διαδίκτυο. Μα είναι η ίδια υποδομή η οποία χωρίζεται, ένα μέρος επιφυλάσσεται για τις managed services και ένα άλλο μέρος επιφυλάσσεται για το ανοιχτό διαδίκτυο. Άρα εμπεριέχεται η σύγκρουση αυτή, αν θέλετε, από την φύση των πραγμάτων. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι στην πρόταση της Κομισιόν αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφέστερο. Έννοιες επίσης όπως recurring είναι ασαφείς νομικοί όροι οι οποίοι δεν ορίζονται σαφώς στην πρόταση κανονισμού και γι' αυτό εμείς ζητούμε να διαγραφούν οι όροι αυτοί από το κείμενο. Συμμεριζόμεθα επίσης τις επιφυλάξεις του συναδέλφου σας της Επιτροπής Περιφερειών. Δεν είναι απόλυτα κατανοητό εφόσον εισάγω νέε ειδικευμένε υπηρεσίες οι οποίες θα οδηγήσουν σε υψηλότερα κέρδη των ε, επιχειρήσεων Telecom Ποιο άραγε κίνητρο θα έχουν οι επιχειρήσεις Telecom να μην πωλήσουν όσο γίνεται περισσότερες από αυτές τις ειδικευμένες υπηρεσίες. Και εδώ λοιπόν εμπεριέχεται το ενδεχόμενο σύγκρουσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν οι ειδικευμένες υπηρεσίες. Νομίζουμε όμως, και εδώ πρέπει να εγκύψουμε λίγο και στη βασική ιδέα των προτάσεων της Κομισιόν, η εντύπωση που έχουμε εμείς από την ανάγνωση του κειμένου της Κομισιόν είναι ότι πρέπει να καταγράψει τις δυνατότητες εισαγωγής ειδικευμένων υπηρεσιών και μετά έρχεται η διασφάλιση του ανοιχτού, του, του ανοιχτού διαδικτύου. Έτσι γίνεται στο κείμενο της Κομισιόν. Εμείς θα θέλαμε να το δούμε διαφορετικά, ότι ο κανονισμός εξασφαλίζει πρωτίστως το ανοιχτό διαδίκτυο και μετά δίνει τη δυνατότητα ειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες εν μέρει ήδη υπάρχουν. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Απευθύνομαι στην κυρία Δελκαστήγιο. Η, σύγκρουση, η σύγκριση μάλλον με τους δρόμους είναι επιτυχημένη. ειδικά όμως από την σκοπιά των μίντια θα προσπαθήσω να την κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Όπως είχα πει ήδη προηγουμένως, για μας το διαδίκτυο πρωτίστως είναι πλατφόρμα επικοινωνίας και τρόπος και μέσων παροχής πληροφοριών ή συλλογής πληροφοριών ή ε, αναζήτησης καλύτερα πληροφοριών από την πλευρά των πολιτών, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν άποψη βασισμένη σε διάφορες απόψεις άλλων. Γι' αυτό θεωρούμε ότι βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που πιστεύουν τα μέσα είναι ότι αυτό δεν αρκεί. Στον κανονισμό περί μέσων ενημέρωσης αναγράφεται κιόλας ότι πρέπει εκ των προτέρων να αποκλείονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, υπάρχει μια σφαλμένη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολο να, γίνει, να αντιστραφεί. Πάλι εδώ έρχομαι στο παράδειγμα σας με τους δρόμους. Υπάρχουν στους δρόμους πολλοί κανόνες οι οποίοι ε, εξυπηρετούν όσο γίνεται να μειωθεί ο κίνδυνος ένα αυτοκίνητο να χτυπήσει ένα πεζό. Έχουμε σήματα, έχουμε φωτεινούς σηματοδότες, περιορισμούς ταχύτητας, δηλαδή έχουμε μια ολόκληρη σειρά κανόνων που αποσκοπούν στην πρόληψη. Δεν λέω ότι χρειαζόμαστε κώδικα οδικής κυκλοφορίας για το διαδίκτυο, ασφαλώς όχι. Αλλά νομίζω ότι από την σκοπιά μας μπορώ να πω ότι είναι σημαντικό μέσα σε όλες αυτές τις ευκαιρίες που ανοίγονται να διακρίνουμε και τους ενδεχόμενους κινδύνους και τουλάχιστον να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις που να έχουν και προληπτικό χαρακτήρα ή τουλάχιστον να μπορούμε να αντιδρούμε ταχύτατα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις ε, και σε σχέση με αυτό που είπατε θα ήθελα να πω δύο λόγια. Το ίντερνετ είναι ε, μια τρομερή πλατφόρμα επικοινωνίας, είναι μια πλατφόρμα η οποία ε, επιτρέπει την επικοινωνία βεβαίως είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει παγκόσμια διάσταση. Ωστόσο, το ίντερνετ θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των επιχειρήσεων. Ε, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αγορές. Ε, μας δίνει τη δυνατότητα να, μάλλον και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο εργαλείο εξαιρετικά ε, ευρύ ε, το οποίο ξεπερνάει την επικοινωνία. Επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας που γίνεται εκτός του ίντερνετ. Επομένως, σας αποφύγουμε να δημιουργήσουμε μία εικόνα του ίντερνετ μονοδιάστατη θα πρέπει το ε, ίντερνετ να χρησιμοποιήσει το δυναμικό του έτσι ώστε να έχει επίπτωση στην ε, οικονομική ανάπτυξη και θα το πούμε, θα το ξαναπούμε, θα το επαναλάβουμε ad ότι ε, integradora y no excluyente y ε, μέχρι ότου κατανοήσουν όλοι ότι η προσέγγιση προς το ε, ίντερνετ δεν θα πρέπει να είναι συσταλτική ε, και ούτε να περιορίζεται μονάχα στον τομέα της επικοινωνίας. Αυτό θα αποτελέσει πολύ μεγάλο σφάλμα ε, κατά αυτή την έννοια λοιπόν και κατά την άποψή μου θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να δώσουμε ε, στο ε, διαδίκτυο αυτήν την δυνατότητα ακριβώς να συμπεριλάβει πολλούς, πολλές δραστηριότητες και ε, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και τους μηχανισμούς αυτούς που θα μας επιτρέψουν ε, μέσω σαφών διεργασιών ε, να μπορούμε και να ελέγχουμε. Ακριβώς επειδή το ίντερνετ είναι ένα τόσο διευρυμένο εργαλείο. Επαναλαμβάνω πάντως ότι ο πυρήνας του διαδικτύου πρέπει να είναι ένας πυρήνας ολοκληρωμένος και όχι ένας πυρήνας αποκλεισμών και όλοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ε, να ε, χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Επίσης, Είχατε, μου είχατε απευθύνει και μια ερώτηση προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με την ε, τροπολογία μου για διαγραφή του άρθρου 19. Ε, κοιτάξτε, τώρα θα αρχίσει το δεύτερο πάνελ και θα σας κάνω στα πλαίσια αυτής, ε, αυτού του δεύτερου πάνελ, θα σας απαντήσω στο θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν τώρα το δεύτερο πάνελ, το οποίο αφορά την ενιαία αδειοδότηση για τη λειτουργία σε διάφορες χώρες μέλη, ε, προϊόντα πρόσβασης και μπέρεκ. Ευρωπαϊκός ε, φορέας ε, λοιπόν, θα δώσω μάλιστα τον λόγο αμέσω στον πρόεδρο του Μπέρεκ, τον δόκτωρα Λεωνίδα Κανέλο. Μετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λουίτζι Γκαμπαρντέλα ε, της ΕΤΝΟ και μετά στον Άντριαν Whitchurch, αντιπρόεδρο για ευρωπαϊκά θέματα ε, της British Telecom, του ομίλου British Telecom. Θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του Μπέρεκ, τον δόκτωρα Λεωνίδα Κανέλο. Dear uh, members. Κυρία Σαρτόρη, κυρία Πιλάρ Νταλκαστίγιου, μέλη της Επιτροπής Ήτρε, κυρίες και κύριοι. Ως πρόεδρος της ΜΠΕΡΕΚ, το Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις ε, ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες, να σας ευχαριστήσω εσάς και να, να χαιρετήσω και τους υπόλοιπους παρεμβαίνοντες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την ακρόαση. Θέλουμε να υπάρχει μια σωστή αρχιτεκτονική στη ρύθμιση του διαδικτύου. Γι' αυτό υπάρχει το σώμα μας και προσπαθούμε να συντονίσουμε τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την έγκριση του κανονισμού Μπέρεκ το 2009. Είμαι βέβαιος ότι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε τη δήλωσή μας στις 16 Σεπτεμβρίου μαζί με την συνοπτική θέση μας της 17ης Οκτωβρίου 2013. Εκεί εκφράσαμε την ε, άποψή μας για τους υψηλούς πολιτικούς στόχους που υπονοεί το ε, πρόσφατο πακέτο, δηλαδή να προωθηθεί η ενιαία αγορά για τις ηλεκτρονικές ε, τηλεπικοινωνίες και να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες για το όφελο των Ευρωπαίων καταναλωτών και συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Στην παρουσίασή μου, σύντομα, θα αναφέρω τα τρία στοιχεία που θα μας απασχολήσουν στην παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα η νέα διαδικασία διοδότησης, δεύτερον ε, η πρόσβαση και οι δυνατότητες ένδικων μέσων και μετά η διακυβέρνηση. Η Μπέρεκ στην συνοπτική θέση της 17 Σεπτεμβρίου, ε, Οκτωβρίου συγγνώμη, μίλησε για την ανάγκη να ε, εξελιχθούν τα παράλογα ε, εμπόδια στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φορέας μας επίσης εξέφρασε την άποψή του και την πεποίθησή του ότι ένας τέτοιο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με μια ενιαία προσέγγιση που διασφαλίζει και την προβλεψιμότητα και την νομική βεβαιότητα. Προκειμένου να επιδιώξουμε αυτό το σκοπό πρέπει να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση του ίδιου template και αυτό το επιδιώκει με το έργο της ε, η Μπέρεκ. Μία ενιαία ε, κοινοποίηση και αδειοδότηση θα πετύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ ενός, ενός καθεστώτος light για την αδειοδότηση που θα διευκολύνει τους προμηθευτές και από την άλλη την ανάγκη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να διασφαλίσουν τη σωστή εποπτεία της αγοράς. Βάσει αυτών των στοιχείων μπορούμε τους ερχόμενους μήνες να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την πρόταση η οποία συνάδει με τις βασικές ιδέες που εκφράζονται και στο σχέδιο έκθεση της Επιτροπής Ήτρα. Συγκεκριμένα μπορούμε να εντοπίσουμε τις λεπτομέρειες μιας προηγμένης διαδικασίας αδειοδότησης μαζί με το ενίο έντυπο για την ε, κοινοποίηση. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε και λεπτομερή πρόταση μέσα στο 2014 ώστε να επιταχυνθεί η όλη νομοθετική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πρόσβασης και τα ένδικα μέσα, αυτό έχει να κάνει με την προσέγγιση που θα επιλέξουμε εφόσον υπάρξει προτίμηση για συγκεκριμένη, συγκεκριμένα ένδικα μέσα ε, στην αγορά. Νομίζουμε η καλύτερη επιλογή θα είναι αυτή που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στο τοπίο του διαδικτύου, στις τεχνολογικές λύσεις που προτείνονται και στις διαφορετικές ανάγκες ανά την Ευρώπη. Αυτά ε, συνεχώς μεταβάλλονται με το χρόνο ούτως ή άλλως. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την επιλογή που έγινε στο σχέδιο έκθεση τη ΣΥΤΡΕ. Η Μπέρεκ θέλει επίσης να προτείνει το να δημιουργηθούν ε, προσεγγίσεις βάσει των βέλτιστων ρυθμιστικών ε, πρακτικών για τα ε, προϊόντα χοντρικής στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι θα διευκολύνουμε και τι εταιρείε και του καταναλωτέ, ώστε να ξέρουν ότι τα προϊόντα αυτά διαρκώ ε, ενημερώνονται, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τι εξελίξει στην αγορά. Ω προ την ίδια την ε, Μπέρεκ, θεωρούμε ότι η θεσμική τη διοργάνωση πολύ σωστά έχει σχεδιαστεί, ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργική τη ανεξαρτησία. Οποιεδήποτε αλλαγέ επέλθουν προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία τη Μπέρεκ, θα πρέπει να γίνουν με κάθε δυνατή επιφύλαξη, διότι μην ξεχνάμε και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που θα αποτιμήσει το έργο του Μπέρεκ. Πρέπει να υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο πρακτικών για την Μπέρεκ, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητά μας να ε, διαδραματίσουμε σωστά το ρόλο μας. Μία τέτοια πρόνοια θα επιτρέψει και θα διευκολυνθεί μάλλον από την απλουστευμένη διαδικασία διοδότηση. Προαπέτηση βέβαια για να λειτουργήσει εύρυθμα μια τέτοια διαδικασία είναι οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ να λάβουν την αρμοδιότητα βάσει νομοθεσία, να έχουν ε, τι δυνατότητε αδειοδότηση. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώ και πρέπει να το πω αυτό από τη θέση μου. Να κλείσω τη σύντομη μιλία μου, εκφράζοντα την ε, επιθυμία τη ΜΠΕΡΕΚ να συνεργαστεί στενά με όλου του θεσμικού ε, ενδιαφερομένου, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια τελική πρόταση κανονισμού που θα ε, εξυπηρετήσει του μακροπρόθεσμου σκοπού μα χωρί να υπονομεύει τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Πλαισίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Eh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κανέλο, πρόεδρε του Μπέρεκ. Το λόγο έχει ο κύριος Λουίτζι Γκαμπαρντέλα, πρόεδρος της ΕΤΝΟ. Αγαπητή πρόεδρε. Αγαπητή Πρόεδρε, κυρία Μαρία Σαλτώνη, κυρία εισηγήτρια Πιλάρντε Καστίγιο, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις μου σε αυτήν την τόσο σωστή χρονική στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το σώμα που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες, άρα είναι το σπίτι μας. Και η θέση του Κοινοβουλίου πάνω στα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι προαλήσαντες ε, ε, εκφράσαν τις απόψεις μας, ε, σχετικά, τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να αρθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες. χρειαζόμαστε ε, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και εδώ θα συμφωνήσουμε με τον πρόεδρο του Μπέρεκ, τον φίλο μου κύριο Κανέλο, αλλά βεβαίως ε, και ίσους όρους ε, ανταγωνισμού. έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε αυτήν την, ε, ε, ε, την αντιπροσωπευτική θέση όσο και αν αλλάξει η νομοθεσία. Θα πρέπει τούτη τη στιγμή να προσαρμόσουμε την νομοθεσία στην αγορά που πλέον έχει αλλάξει και δεν, ισχύει, δεν ισχύουν πλέον εδώ οι όροι που ίσχυαν 15 χρόνια πριν. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν σωστά οι σε προκλήσεις. Οι συνθήκες πλαίσιο πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε να ε, ε, εποφεληθούν ε, και οι ε, πολίτες ε, που είναι και χρήστες. Κατά αυτήν την έννοια η ΕΤΝΟ λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις κινήσεις του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παραγάγει πολύ σωστά αποτελέσματα τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τους Ευρωπαίους πολίτες έχουν ξεκινήσει βήματα προς αυτήν την ε, κατεύθυνση, κυρίως ε, με την έκθεση για την πολιτική του φάσματος. Ε, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια κυρία Πιλάρτε Καστίγιο γιατί κατά την άποψή μας ε, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αρθεί ε, η ασάφεια και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε νομική σαφήνεια. Η Ευρώπη πρέπει και οφείλει να είναι περισσότερο φιλόδοξη. Η πρόταση του κανονισμού θα πρέπει να δοθεί σαν ένα εργαλείο Ε, Ο συνομοθέτη μπορεί να κάνει τη διαφορά έτσι ώστε η δέσμη αυτή να βελτιώσει ακόμα περισσότερο και να διευκολύνει τις περαιτέρω επενδύσεις ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει τις σωστές επιλογές, αυτές δηλαδή οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ε, επενδύσεων θετικό ε, και προς τον χρήστη. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες σκέψεις. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, η υψηλή ε, συνδεσιμότητα είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Ε, και εδώ σχετίζονται και θέματα όπως η ευφυής, the smart grids, καθώς επίσης και άλλα θέματα όπως είναι το υπολογιστικό νέφος κτλ. Ε, ε, ε, εμείς θεωρούμε ότι στην έκθεση η οποία μας έχει υποβληθεί δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση των τηλεπικοινιών σε συμβατικούς όρους μειώνεται 2% κάθε χρόνο. Ε, η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λόγω και της παρουσίας πολλών παρόχων αλλά και λόγω μεγάλων Ιντερνετικών ε, εταιριών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μια σαφή, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ε, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι νέες ε, ικανότητες, οι νέες υποδομές μάλλον οι οποίες θα στηρίζουν τις ικανότητες της συνδεσιμότητας. Δεν θα πρέπει η ρύθμιση να είναι κάτι ανασχετικό ε, απλώς. Μέσω της ρύθμισης θα πρέπει και η καλύτερη πρόσβαση να διασφαλίζεται, αλλά και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι ένα πραγματικά ε, ίσο πεδίο για όλους λείπει ακόμα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον Ευρωπαίο καταναλωτή χωρίς κανένα δίκαιο ε, ε, όταν μιλάμε για κοινωνικές πλατφόρμες, ε, για παρόχους επικοινωνίας στο ίντερνετ, λοιπές πλατφόρμες applications κτλ. Μεγάλη διαφάνεια χρειάζεται, καμία διακριτική μεταχείριση, φορητότητα, ε, δικαιώματα τα οποία ε, μπορούν να εφαρμοστούν ε, και για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου σε αυτήν την συγκλίνουσα αγορά. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικοί παίχτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια όσον αφορά την διασύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Μπέρεκ η αλλαγή, η τροποποίηση της παρούσας αρχιτεκτονικής θα πρέπει να βασίζεται στην λογοδοσία. Η ε, αλληλενέργεια ανάμεσα στον Μπέρεκ, την Κομισιόν και την αγορά ε, θα πρέπει να μην δημιουργήσει με κανένα τρόπο ρυθμιστική ασφάλεια, ασάφεια. Συγγνώμη. Είναι το τελευταίο που θέλουμε αυτή η ρυθμιστική ασάφεια και επίσης θα πρέπει να αποφευχθεί ε, η στρέβλωση της αγοράς ε, θα, ε, η ρυθμιστική ε, μια ελλειπής ρυθμιστική κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη στερεύλωση στην αγορά. Ας το αποφύγουμε αυτό. Θα πρέπει όμως να να δράξουμε την ευκαιρία αυτή έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κανόνες τέτοιους τόσο σαφείς ε, και τόσο συγκεκριμένους που θα ανοίξουν το δρόμο σε επενδύσεις ε, στον τομέα αυτό. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Η αγορά χρειάζεται οπωσδήποτε τέτοιου είδους επενδύσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Καστίγιο. Κύριε Βιτ Church. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε και εσείς τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Γνωρίζω ότι δεν κάνανε τόσους πηχαίους τίτλους τα προϊόντα Access όπως άλλα, αλλά εμείς τα βρίσκουμε πολύ σημαντικά και θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί η BT είναι υπέρ ορισμένων των μέτρων που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προτάσεις. Ως εισαγωγικό μέρος πρώτα, η BT εξυπηρετεί πελάτες σε πάνω από 170 χώρες του κόσμου κατορθώνουμε να επενδύουμε άλλωστε πολλά δισεκατομμύρια σε δίκτυα ινών, οπτικών ινών και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επίσης και σε δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων. Πέραν δε του Ηνωμένου Βασιλείου, το βασικό έργο της επιχειρήσεώς μας είναι οι προσφορές υπηρεσιών και στην Ευρώπη και στον κόσμο και γι' αυτό για μένα το βασικό στοιχείο των προτάσεων της Επιτροπής είναι η πρόσβαση. Τώρα γιατί είδους, γιατί είδους πελάτες μιλούμε πέραν των εθνικών συνόρων. Εμείς στοχεύουμε ιδίως σε multi-sites και multinational και corporate customers, δηλαδή εταιρείες κλπ. Δεν μπορείτε να τα διαβάσετε βέβαια, είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Σας δείχνει όμως, σας δίνει μια εικόνα όμως της περιπλοκότητας. Ορισμένοι πελάτες ζητούν υψηλή ανθεκτικότητα του δικτύου, υψηλές ταχύτητες και ούτω καθεξής. Αυτοί οι πελάτες, οι άλλοι τώρα απέναντι στους καταναλωτές, είναι λίγοι σε αριθμό, έχουν όμως 40% της απασχόλησης και 50% του κύκλου και βρίσκουν ε, σημαντικό να έχουν έναν ενιαίο πανευρωπαϊκό πάροχο για να τους εξυπηρετεί. Γιατί τώρα να μην είναι το αντίθετο ε, μια καλή επιλογή. Βλέπετε εδώ ένα είδος φωτογραφίας της ποικιλία των διαφορετικών ρυθμιστικών των διαφορετικών ρυθμίσεων, των διαφορετικών προϊόντων και επαγνωρίζω ότι έχει επικριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένους κύκλους επειδή δεν, έχουν, δεν έχει υποβάλει αρκετά στοιχεία για το πρόβλημα. Αλλά εδώ βλέπετε ότι προβάλλονται τα στοιχεία αυτά και η ασυνέπεια που προκαλείται οδηγεί σε έλλειψη αποδοτικότητας αυξάνει τα βάρη τελών εισφορών κλπ. Σε, ολόκληρο, σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε βάρος των πελατών και των τελικών χρηστών. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Οι προτάσεις απλοποίησης των αδειοδοτήσεων μπορούν να βοηθήσουν. Αν και δεν νομίζουμε εμείς ότι αυτό είναι το βασικός φραγμός για την είσοδο. Πιο πολύ είναι η νομοθεσία περί ε, πρόσβασης. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρώτα προϊόντα πρόσβασης που να είναι fit for purpose, κατάλληλα για το σκοπό που εξυπηρετούν. Επίσης, χοντρική πρόσβαση σε Ethernet. Διαφάνεια, μη διάκριση κλπ από άποψη ρυθμιστική δηλαδή. Επίσης συνέπει και συνεκτικότητα στις χώρες μέλη διότι παρόλο που αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της ΜΠΕΡΕΚ, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου να προβλέψουν κάποια εναρμόνιση αλλά 28 χώρες μέλη ασφαλώς οδηγούν σε μια κατακαιρματισμένη αγορά. Εμείς ε, αναζητούμε συνεκτικότητα στην προσέγγιση και είναι σωστό να σημειώσουμε ακόμη ότι όταν κανείς παρέχει υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκή βάση, είναι αδύνατο να κάνει οικονομίες κλίμακος με την πρόσβαση που προσφέρει παντού. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Όσον αφορά τα εικονικά προϊόντα και τις προτάσεις που καταθέτει η Επιτροπή διότι η φυσική πρόσβαση δεν θα είναι πάντοτε επιλογή, η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι επίσης σημαντική. Κατανοούμε γιατί η Μπερέκ και άλλοι αντιτίθενται σε κάποια κατεύθυνση που θα λέει ότι πρέπει να δώσετε προτεραιότητα σε αυτά απέναντι στα φυσικά προϊόντα. Αυτό που θεωρούμε όμως εμείς είναι ότι ο ρυθμιστής πρέπει πάντοτε να εξετάζει και προϊόντα virtual access, εικονικής πρόσβασης περισσότερο από ό,τι το πράττει για την ώρα. Εν συνόψη λοιπόν υποστηρίζουμε κατ' ουσίαν τις προτάσεις της ε, Κομισιόν ιδίω για την Ethernet Access θεωρούμε ότι μπορούν να βελτιωθούν οι προτάσεις καλύτερα αυτό παρά να ανατραπούν εντελώ. θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταδείξει την ανάγκη για ανάληψη δράσης στο επόμενο νομοθετικό πλαίσιο, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες πανευρωπαϊκά για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας και σε οικονομική ανάπτυξη. Τα οικονομικά ωφελήματα μπορούν να ανέφθουν και σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις είναι αυτές, αλλά σας δίνουν περίπου μια ιδέα της αξίας που μπορεί να δημιουργηθεί. Να ξεκινήσουμε τώρα με τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ξεκινάμε με τους συναδέλφους βουλευτές, μετά έχουμε και τους εκπροσώπους της Επιτροπής των ε, Περιφερειών. Η κυρία Τροκμάν, ευχαριστώ πολύ Πιλάρ για την ενιαία διαδότηση θα είμαι σύντομη διότι δεν ε, συνείδησα κανέναν κατά τις διαβουλεύσεις που να στήριξε την πρόταση ως έχει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως ε, άκουσα να μιλάνε πολύ για περιτά στοιχεία ή για ε, επιπλοκές, περίπλοκες διατυπώσεις. Η απλούστευση λοιπόν νομίζω ότι είναι μια κατεύθυνση που όλους θα μας βρει σύμφωνος. Απλούστευση και ε, αναζήτηση μια συγκεκριμένη ε, ρεαλιστική μορφή διοργάνωση. Ω προ τα υπόλοιπα εναρμονισμένα προϊόντα πρόσβαση, καταλαβαίνω ότι κάποιε προτάσει μπορεί να είναι ενδιαφέρουσε, ε, κάποιε φορέ είναι και η μόνη επιλογή εκτό από ελκυστικέ, αλλά αυτέ είναι η εξαίρεση. Δεν κατανοώ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να γενικεύσει σε τέτοιο βαθμό αυτήν την λύση για να γίνει μια λύση συστηματική. Γιατί εφόσον αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήδη από τους εθνικούς ρυθμιστές, αυτοί είναι ουσιαστικά οι δικαστές, γιατί αυτή η διπλή δυσκολία να περιοριστεί το περιθώριο λιγμών των εθνικών ρυθμιστών και να αποσταλεί ένα αρνητικό μήνυμα, ιδίω για την κλίμακα των επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά το Μπερέκ, την Μπερέκ. Εγώ συνεργάστηκα με τον ε, συνάδελφο Ζαντό για την έκθεσή του που εξετάστηκε ήδη και ψηφίστηκε στην Ολομέλεια. Έκθεση που νομίζω πετυχαίνει μια σωστή ισορροπία. Νομίζω λοιπόν για σκοπούς διακυβέρνησης, ναι, βελτίωση μπορεί να υπάρξει, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με την εισηγήτριά μας, την Πιλάρ Καστίγιο. η Προεδρία μπορεί να οριστεί μεταξύ των μελών και η θητεία μπορεί να εξεταστεί ως προς τη διάρκεια της. Όμως η αρχική πρόταση δεν είναι αποδεκτή εφόσον θέλουμε να είναι ανεξάρτητο το ΜΠΕΡΕΚ ε, έναντι των εθνικών ρυθμιστών ή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Νομίζω λοιπόν ότι η σκοπιά του Ευρωκοινοβουλίου όπως μας φάνηκε και στη συζήτηση που έγινε, είναι πιο ε, εύστοχη. Και θα ήθελα την άποψη και των συμμετεχόντων για τα θέματα αυτά. Κάποιος άλλος συνάδελφος. Γιατί μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις από το κοινό, εάν έχουμε χρόνο. Άλλες ερωτήσεις από συναδέλφους. Ήθελα και εγώ να πω κάτι στη φάση αυτή, διότι οι δικές μου προτάσεις διαφέρουν ελαφρώς από τις προτάσεις του κειμένου της Επιτροπής για αυτό που είπε η κυρία Τροτμάν, συνάδελφος. Πρότασή μας είναι να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία του Μπερέκ Ε, αλλά το θέμα είναι τι επιλογή θα κάνει η Επιτροπή. θα επιλέξουμε μέτρα για να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση εντός του Μπερέκ. Οι εθνικοί ρυθμιστές θα επιλέξουν ε, αρμοδιότητες που είναι κοινέ θα υπάρχει ομοιομορφία ή ασυμμετρική διοργάνωση εφόσον όλοι οι ρυθμιστές δεν έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες στο κάτω τους. Και ως προς τα προϊόντα πρόσβασης, ιδιαίτερως για το διαδίκτυο, Ε, για, τα, για την κυρία Τροτμάν να πω Είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι και οι οργανώσει που επηρεάστηκαν από αυτό το σημείο και επέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι η προτεραιότητα δίνεται σε προϊόντα που δεν καλύπτουν αναγκαστικά τις περισσότερες ανάγκες των χρηστών σε εθνικό επίπεδο. Και κατά δεύτερον, μιλάμε για μια πρόταση, για μια πρωτοβουλία μάλλον, η οποία δεν προκάλεσε αρκετή συζήτηση, δεν εξετάστηκε αρκετά. και δεν υπήρξαν αρκετέ δημόσιε διαβουλεύσει για να συνδυαστούν διαφορετικέ απόψει. Η πρόταση λοιπόν δεν είναι αρκετά όρημη. Εγώ πρότεινα να διαγραφεί το άρθρο και οι διατάξεις για τα προϊόντα πρόσβασης στο ίντερνετ. Α, αλλά γιατί μου φάνηκε πιο αναγκαίο να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τις γνώσεις που είναι διαθέσιμες για το πώς θα εξορροπήσουμε τη ζήτηση με την προσφορά. Ίσως έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα σε διαφορετικά προϊόντα. De comunicaciones electrónicas, que por cierto he propuesto una fecha. Υπάρχει και η οδηγία για τις τηλεπικοινωνίες, ασχολούμαστε και με την αναθεώρησή της, αλλά τον Ιούλιο του 2016 eh, ίσως να τα ξαναδούμε αυτά ως μέρος αυτής της διαδικασίας αναθεώρησης. Καταλαβαίνω λοιπόν και την συλλογιστική του εκπροσώπου της British Telecoms Business to business είναι η προτεραιότητά σας. Έχετε συγκεκριμένες επιλογές όταν μιλάμε για προϊόντα πρόσβασης. Όμως, το πρόβλημα είναι ποιος είναι ο συνομιλητής σας συνήθως. Λίγοι είναι αυτοί που αντέδρασαν σε θετικά, θετικά στα προϊόντα πρόσβασης. Όλοι βλέπουν το θέμα από τη δική τους σκοπιά el sector o para el país, dependiendo de eh, qué instituto. Que... Άρα το θέμα είναι ότι είναι πιο κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο τομέα, για μια συγκεκριμένη χώρα. Ε, τα πάντα εξαρτώνται από τον ε, τομέα εργασίας του καθενός. Εγώ λοιπόν κάπως ε, πρέπει να πω ότι αισθάνομαι δυσαρέσκεια θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και για τα θέματα αυτά σε κάποια φάση. Ιδάλω, θα παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση. Ο καθένα να υποστηρίζει το δικό του. Νομίζω θα άξιζε τον κόπο να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό, να δούμε πώς η εναρμόνιση μπορεί να προσφέρει κάτι. Por tanto, lo que me ha parecido más oportuno, y está sujeto naturalmente a que lo discutamos en el Parlamento, es eh, posponerlo, posponerlo a un debate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 ε, ε, και θα πρέπει αυτό να γίνει με τρόπο που να είναι αποτελεσματικό. Η αρχική πρόταση ήταν πολύ περίπλοκη. Θεωρούμε όμως ότι το Κοινοβούλιο έχει υποχρέωση να προσπαθήσει να απλουστεύσει Βλέπω ότι δεν υπήρξαν ε, ερωτήσεις, αλλά ήθελα να δώσω την ευκαιρία στους ε, συμμετέχοντες να κάνουν κάποιο επιπλέον σχόλιο, αν το θεωρούν σκόπιμο. Παρακαλώ. Εγώ προσωπικά πρέπει να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Τροτμάνα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να επανέλθουμε στην θέση του Μπέρεκ, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ σαφής. Βεβαίως ε, πιστεύουμε ότι η ύπαρξη απλουστευμένου ε, εντύπου οπωσδήποτε θα απλουστεύσει για το σύστημα, επομένως ε, εφαρμόζουμε την αρχή ότι αν κάτι λειτουργεί δεν χρειάζεται να το αλλάξεις, να το χαλάσει Περιμένουμε λοιπόν, ε, προτιμούμε συγγνώμη αυτήν την ε, πιο ε, απλού, απλή προσέγγιση. Όσον αφορά την πρόσβαση σε εναρμονισμένα προϊόντα, το ΜΠΕΡΕΚ θέλει να διασφαλίσει το δικαίωμα των operators να παρέχουν ποιοτικά προϊόντα, αλλά ε, δεν συμφωνούμε με τις προκατασκευασμένες λύσεις. Η ευελιξία λοιπόν, ε, η ευελιξία και η δυνατότητα ε, προσαρμογής των προϊόντων, στην, των προσφερόμενων προϊόντων στις διαφορετικές αγοράς, αγορές, με όποιες διαφορές ή ιδιαιτερότητες έχουν οι αγορές αυτές, είναι κάτι σημαντικό για μας. Δεν έχουμε βεβαίως αποδείξεις ε, ε, σχετικά με λήψεις ε, στην αγορά οι οποίες θα οδηγήσουν στην εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων remedies ε, μέτρων διόρθωσης αλλά πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε εκ των προτέρων ε, και τα τεχνικά και τα νομοθετικά εργαλεία έτσι ώστε όταν παρουσιαστεί ανάγκη να μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης το Μπέρεκ οπωσδήποτε συμφωνεί με την ε, διάδοση συγκεκριμένων βελτίστων πρακτικών. Τελευταίο σημείο λοιπόν το οποίο σχετίζεται και με την διακυβέρνηση του Μπέρεκ Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του Μπέρεκ απέναντι και στους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και απέναντι στις εθνικές μυστικές αρχές. Όσον αφορά τώρα την πρότασή σας για την επιλογή του εκτελεστικού διευθυντή της Μπέρεκ, ο οποίος θα επιλεγεί από τα μέλη ε, θεωρούμε ότι η πρόταση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και σας διαβεβαιώ ότι στην ε, ολομέλεια της, ε, του οργάνου μας την επόμενη εβδομάδα σε Βουδαπέστη θα μεταφέρουμε αυτό το θέμα στους συναδέλφους. Πολύ ωραία, εδώ έχουμε δύο συμμετέχονται στο επόμενο πάνελ που θέλουν να παρέμβουν και να υποβάλουν ερωτήσεις. Λοιπόν, να δείξουμε κάποια ευελιξία, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλέ ερωτήσει από πλευρά των Ευρωπαίων βουλευτών. και στο τέλος βέβαια, αν έχουμε χρόνο, θα ξεκινήσουμε, θα ανοίξω ένα γενικότερο πάνελ ερωτήσεων έτσι ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει όλες τις ιδέες του και τις απόψεις του. Πολύ σύντομα θα σας δώσω τον λόγο όσον αφορά τα προϊόντα πρόσβασης και μετά θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ο κύριος Γκαμπαρντέλα από το προηγούμενο πάνελ ήθελε να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα νομίζω ότι είναι σημαντικό, κάτι που είπα και προηγουμένως και θέλω να το επαναλάβω. Εμείς είμαστε στρατευμένοι, έχουμε αποφασίσει απόλυτα να συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εάν μπορούν να βρεθούν συμβαστικές λύσεις, ε, βεβαίως θα τις ε, μελετήσουμε πολύ θετικά. Αλλά ας δούμε τι είναι σημαντικό για μας. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Είπατε τη μαγική λέξη απλούστευση. Δεν μπορούμε να απλουστεύσουμε εάν δημιουργήσουμε κι άλλους κανόνες. Όσον αφορά την ενιαία ε, αδειοδότηση, την πρόσβαση στο φάσμα κτλ το σύστημά μας, το ευρωπαϊκό σύστημα είναι πολύ μπερδεμένο. Είναι το πιο περίπλοκο σύστημα ε, στον κόσμο. Και εν παρόδο να πω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, ε, η, πιο, ε, είναι η περιφέρεια του κόσμου με την περισσότερη νομοθεσία. Επομένως χρειαζόμαστε απλούστευση. Είναι σημαντικό και για τις εταιρείες, είναι σημαντικό και για τους ρυθμιστές. Προφανώς υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι θετικά. Εδώ έχουμε μια σύσταση ε, πολύ σημαντική, η οποία είναι μετά από ε, δύο χρόνια όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών του χαλκού και για τις ίνες. Ε, αυτή η σύσταση, αυτές οι σύστασεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να τις δούμε από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο ερωτήσεις σύντομες από την κυρία Φιτόρη και από τον κύριο Μάρκους της WIC και της ΕΚΤΑ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να σχολιάσω τα ε, γενικά προϊόντα πρόσβασης και την ενιαία εξουσιοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι το ισχύον ρυθμιστικό πρότυπο που βασίζεται στο προκύπτει από το ευρωπαϊκό πλώσιο δίνει τα βέλτιστα δυνατά ωφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές συνολικά. Υπάρχουν ε, πολλές επενδύσεις και σε άλλα μέρη του κόσμου και εκεί μπορεί να βλέπετε μεγαλύτερες δαπάνες από την πλευρά του κεφαλαίου αλλά όχι μεγαλύτερες και περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα. Τίνουν να επενδύουν σε άλλου είδους ε, ε, επιδοτήσεις λόγου χάρη οι ε, εταιρείε και όχι στην κινητή τηλεφωνία λόγου χάρη όπως εμείς. Ένας φορέας τώρα όπως ο ITU ή ο ΣΑΜ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσπαθούν να αυξήσουν τις ταχύτητες, να, γίνουν, να φέρουν σε χαμηλότερα επίπεδα τις τιμές, να γίνουν καλύτερες προσφορές προς τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν περισσότερη πρόσβαση στο ευρωζωνικό διαδίκτυο από ό,τι στις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία και αλλού σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Οπότε είναι ύψη τη σημασία να διατηρηθεί αυτό ο ρυθμό και να βασιστούμε στο τόσο καλά οικοδομημένο ρυθμιστικό μα πλαίσιο. Κάτι που να μα επιτρέψει να βασιστούμε σε αρχέ τη αγορά που να είναι. να μας προετοιμάζουν για το μέλλον, να προλυαίνουν το έδαφος. Για την ευρυζωνικότητα επίσης θα πρέπει το unbundling να επιλεγεί τελικά και να εφαρμοστεί ώστε να μπορούν και οι προμηθευτές να παράσχουν όλες αυτές τις υπηρεσίες στα δίκτυά τους. Το πρότυπο αυτό το εντόπισε και η μελέτη του Ευρωκοινοβουλίου για την Επιτροπή Ήτρε, ε, με το ίδιο αντικείμενο άλλωστε, και θεώρησε ότι δεν θα αλλάξει η τάση των επενδύσεων από την αλλαγή των παροχών των προμηθευτών. Για το άρθρο 18 λοιπόν του σχεδίου κανονισμού και την αιτιολογική σκέψη 38 είναι πολύ σωστές οι προτάσεις της ε, εισηγήτριας. Συμφωνούμε πάρα πολύ με αυτά που είπε ο εκπρόσωπο τη BT παρόλα αυτά, ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη, ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εναρμόνιση. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, σειρά υπηρεσιών που προτείνουμε στι επιχειρήσει επικοινωνιών, αλλά και το κατά πόσον θα υπάρξει σωστή ιεράρχηση ε, των ε, προσφορών Νομίζουμε ότι η νέα αγορά πραγματικά μπορεί να πυροδοτήσει πολύ περισσότερη οικονομική ε, ανάπτυξη εφόσον αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών σε όλους τους τομείς. Αλλά για μας θα ήταν καλό να διατηρηθεί αυτό που αναφέρεται και στο σχέδιο πρότασης. με τα βασικά προϊόντα που προτείνονται ως λύσεις για εταιρείε. Μιλάμε όμως για συμπληρωματικά προϊόντα που χρειάζονται πέραν των βασικών. Για τους ε, ε, χρήστες από τον κόσμο των ε, εταιριών και τους τελικούς χρήστες. Πάντως πρέπει να διατηρήσουμε τους ελέγχους και να επιδιώξουμε την ισορροπία στην κατανομή αρμοδιοτήτων και πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τη Κεντρική Ρυθμιστική Αρχή και των Εθνικών είναι σωστή. Οπότε θα συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια. Για το καθεστώ τη εξουσιοδότηση, συμφωνούμε με το απλουστευμένο και εναρμονισμένο σύστημα διοδότηση, κάτι που θα μειώσει το γραφειοκρατικό άχθο και οι προτάσει τη ηγέτρια μα βρίσκουν σύμφωνο. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ, ο κύριο Μάρκο. Είμαι διευθυντή του WIK, του Γερμανικού Ερευνητικού Ινστιτούτου, και να σχολιάσω τα θέματα τη αδειοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω, στην, σας, στην πρόταση τη αναφέρει αυτό που και ο μιλητή του πάνελ σχολίασε σωστά. Ότι για τι οικουμενικέ υπηρεσίε και την αδειοδότηση υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό που προτείνει βέβαια η Συγκεντρία του είναι πολύ απλούστερο και πολύ πιο λογικό από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη υπάρχουν όμω ε, διευθετήσει για τι πληρωμέ και εκεί που οι υπηρεσίε αυτέ παρέχονται, οι βέλτιστε πρακτικέ που αναγνωρίζει και η Μπέρεκ είναι ε, αρκετέ. Δεν χρειάζεται να επιβαρυνθούν οι μικροί φορεί. Δεν χρειάζεται να Υπάρχουν σοβαρέ αλλαγέ, αλλά μερικέ μερικές, ε, μικρέ διορθώσει. Ε, τα συγχαρητήριά μου σε όλου του ομιλητέ για τι πολύ εύστοχε παρουσιάσει του. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε επομένω στο επόμενο πάνελ, το τρίτο πάνελ σχετικά με το φάσμα. Θα ξεκινήσουμε με τον Νικόλα Φράγκ, ε, επικεφαλής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, την Νικόλα Φράγκ, από την EBU. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε η European Broadcasting Unit ε, και ε, ε, εκπροσωπούμε τις δημόσια φάσματα στην Ευρώπη και αλλού. Πριν ασχοληθώ με το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, θα ήθελα να δραχθώ της ευκαιρίας να σας υπενθυμίσω τον σημαντικό ρόλο που παίζει για την ραδιοφωνική και λυπή αναμετάδοση το θέμα του φάσματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να, να είμαστε σε θέση να ε, ε, ε, επιτύχουμε σχεδόν καθολική υπηρεσία. Οι τελευταίες στατιστικές του Ευρωβαρόμετρου λένε ότι 46% των σπιτιών για την πληροφόρησή τους ε, έχουν την ε, τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αυτό σημαίνει 238 ε, εκατομμύρια, δηλαδή ένα σημαντικό, ένα σημαντικός αριθμός. Εκπροσωπούμε, 2000, έχουμε αυτή τη στιγμή 2.000 κανάλια τηλεοπτικά και με αυξητική τάση μάλιστα. Ε, βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στα πλαίσια της ε, υπηρεσίας μας ε, έχουμε πολλές διαφορές. 50% περίπου είναι εθνικής εμβέλειας και το άλλο 50% αφορά τοπικά και περιφερειακά κανάλια. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει στην προσεκτική μελέτη του νέου κανονισμού και της νέας δέσμης μέτρων. Αυτό σημαίνει βεβαίω ότι και οι αρχές της δέσμη Telecom θα πρέπει να παραμείνουν παράλλακτα. Όσον αφορά την πολιτική του φάσματος, ε, το Telecom Package λέει ακριβώς, ε, αναφέρει ρητά ότι το φάσμα παρουσιάζει ε, πολλαπλές, παρουσιάζει βάρος και αξία και οικονομική αλλά και πολιτιστική. Υπάρχουν Υπάρχουν βεβαίως στοιχεία τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να, διασφαλιστούν, να διευκρινιστούν συγγνώμη, στον, ε, στο κείμενο προκύπτουν βεβαίως διάφορα σημεία. Πρώτον, ε, ο σημαντικός ρόλος του φάσματος ε, που θα πρέπει να αναγνωριστεί για τηλεοπτική και ραδιοφωνική αναμετάθεση και υπάρχει και μία, ε, θα πρέπει να υπάρξει κάποια τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 17 κατά αυτή την έννοια. Δεύτερο σημείο, και τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραμείνουν αναμεμειγμένοι στη διαδικασία αποφάσεων για την ευρωπαϊκή πολιτική φάσματος. Η απόφαση εναρμονισμένου φάσματος είναι πολιτική και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν εμπλεγμένοι. Τα άρθρα 8 και 9 θα πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο ε, έτσι ώστε να είναι σαφής και η έννοια του ανασμονημένου φάσματος. Κατά την ίδια έννοια είναι σημαντικό να μην ε, υπάρξουν αποφάσεις για ε, περαιτέρω εναρμόνιση του φάσματος πέραν των 8 MHz. Ε, γιατί διαφορετικά ε, θα πρέπει, ε, γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα. Κατά αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι ασφαλμένη η αναφορά στα 700 MHz. Θα πρέπει ε, πριν ε, ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης να ληφθούν υπόψη και να μελετηθούν όλα τα κριτήρια. Όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10, ε, έχουν ληφθεί υπόψη αυτές, αυτά τα κριτήρια από τις εθνικές αρχές. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη την, ή, την παρούσα χρήση των φασμάτων και να μελετήσουν εάν γίνεται αποτελεσματική χρήση των ασυρμάτων ε, ε, του ασύρματου φάσματος ε, εκεί όπου αυτό έχει δοθεί ας πούμε δεν μπορεί να τεκμέρεται ότι το ασύρματο ε, δίκτυο και ε, το ασύρματο φάσμα είναι η καλύτερη απάντηση για μεγαλύτερη συνδεσιμότητα. Δεν ε, αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα. Μπορεί μια σταθερή ζεύξη να δώσει εξίσου καλά αποτελέσματα και να είναι καλύτερη επιλογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 3, 3D ή 4D. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη το κόστος ε, ε, το οποίο προκύπτει από την, ε, από την αποχώρηση κάποιων χρηστών από το φάσμα. Είπα προηγουμένως ότι η πολιτική φάσματος ε, είναι ε, πολιτική απόφαση, αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι και τα τεχνικά σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες προκαλούν παρεμβολές ε, λόγω της ε, ιδιωτικής χρήσης του φάσματος ε, και βεβαίως εκεί θα πρέπει να δοθούν τεχνικές λύσεις. Συνοψίζοντας, οι αρχές ε, που ισχύουν στο, στη δέσμη Telecom θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ε, ισχύσουν, θα πρέπει να, να αναγνωστεί ε, η σημασία του φάσματος, κυρίως η αντιλέωση και το ραδιόφωνο. Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραμείνουν εμπλεγμένα στη διαδικασία και η ε, ε, φυστάμινη χρήση καθώς επίσης και το κόστος του φάσματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τελευταίο σημείο, ε, οι ενδεχόμενες παρεμβολές θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν και να διευθετηθούν. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Λοντάν, αντιπρόεδρος της Deutsche Telekom για την ε, πολιτική φάσματος και τα σχετικά προγράμματα. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω την άποψη και τις παρατηρήσεις μας ό,τι αφορά την πολιτική φάσματος. Η γερμανική Telekom συνολικά υποστηρίζει το σχέδιο οδηγίας της ε, ενιαίας αγοράς για την πολιτική φάσματος. Είναι σημαντικό και για την κινητή τηλεφωνία αλλά και για τους πελάτες μας και για όλους τους πολίτες να ξεπεραστεί ο κατακαιρματισμός της αγοράς της Ευρώπης των 28 και κυρίως ό,τι αφορά την αδειοδότηση για τη χρήση του ευρώ φάσματος. Η κατάσταση όπως έχει σήμερα παρεμποδίζει τις επενδύσεις και η κατακαιρματισμένη υποδομή μειώνει την ε, θέση των Ευρωπαίων ε, παρόχων απέναντι στους ανταγωνιστές τους, για παράδειγμα από τις ΗΠΑ. Η πρόταση είναι ένα πρώτο βήμα για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Για να προχωρήσουμε σε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη, τα άρθρα που έχουν σχέση με την πολιτική φάσματος μπορούν να αποδειχτούν ακόμα πιο φιλόδοξα και να δώσουν ακόμα πιο συγκεκριμένες κατευθείαν γραμμές στα χώρα μέλη. Οι operators όπως η γερμανική Telecom που δραστηριοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις από τις διαφορές των ρυθμίσεων και των διαφόρων διαδικασιών. ο στόχος της διαφάνειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης επιβάλλει στους operator να μην επιβάλλουν διακρίσεις στους α, καταναλωτές και επομένως ασφάλεια επενδύσεων. Συχνά οι δημοπρασίες χρησιμοποιούνται για να ενισχύουν τους εθνικούς προπολογισμούς. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Θα πρέπει δε τα τέλη να καταβάλλονται από του operator όταν θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο, δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζουν να το χρησιμοποιούν. Συμφωνούμε με την πρόταση Ήτρε να εκδίδονται άδειε τουλάχιστον 30 ετών, να μπορεί να γίνεται και μίσθωση του δικτύου για να γίνει πιο αποδοτική η χρήση, ουδετερότητα, επίσης οι κανόνες όμως που έχουν σχέση με την απόδοση της τεχνολογίας για ορισμένα ε, φάσματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Αυτά θα πρέπει να, αποφασίζει, να τα αποφασίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Η Γερμανική Τελεκόμ υποστηρίζει επίσης την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να, επιτρέ... να μειώσει τις... τους ρυθμιστικούς περιορισμούς βέβαια με την, ε, με το σεβασμό των δικαιωμάτων των κατόχων των αδειών. Για την media reception τώρα, ακούσαμε κάτι προηγουμένως γι' αυτό και για την εμφαινόμενη σύγκρουση. Στο μέλλον τα δίκτυα ε, δεδομένων θα παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο και για την λήψη εκπομπών και τα, και δίκτυα θα γίνονται όλο και πιο κινητά. Είναι σημαντικό λοιπόν τα κινητά δίκτυα να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της κυκλοφορίας των δεδομένων. Σχετικά με το, με το φάσμα του 700 MHz πρέπει να προβλεφθεί αυτό. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβολές, αυτό σημαίνει μια χρήση co-primary δεν θα είναι δυνατή. Αυτή η αυτό το φάσμα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί στους ε, operator της κινητής τηλεφωνίας εφόσον υπάρχει τέτοια ζήτηση. Για τη μελλοντική χρήση όμως θα πρέπει να ακούσουμε τους πελάτες και να εκπονήσουμε τα πιο αποδοτικά συστήματα για το μέλλον χωρίς προκαταλήψεις. Εν τέλει, ο κανονισμός που προτείνεται για την ενιαία αγορά είναι καλός και για την αγορά και για τους χρήστες του φάσματος και με κάποιες τροποποιήσεις μπορεί να αποτελέσει επιτυχία για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. And now we have... Ευχαριστούμε πολύ. Και εν τέλει ο κύριος Ποχοχέλ. Καθηγητής Οικονομικών στην Telecom Tech. Uh, Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Να κοιτάξουμε μαζί τη χρήση του ραδιοφάσματος στην Ευρώπη και τους όρους της χρήσης, της αυτής. Έχουν ε, ήδη γίνει πολλά και το Ευρωκοινοβούλιο ιδίως έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση για την πρόσβαση στο, ραδιοφάσμα και η ποικιλία των δράσεων που έχουν ε, βασιστεί στην πρόσβαση στο ραδιοφάσμα είναι μεγάλη. Ωστόσο, εάν δούμε την σημερινή κατάσταση, μου φαίνεται ότι αυτό που στοχεύουμε η ύπαρξη μιας ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη είναι κάτι που δεν το επιδιώκουν επαρκώς οι προτάσεις που τώρα έχουν υποβληθεί. Αληθεύει ότι οι τιμές για την κινητή τηλεφωνία στην Ευρώπη είναι χαμηλές σχετικά. Αυτό είναι πολύ καλό για τους καταναλωτές. Αν δούμε όμως τη συνολική διάρθρωση της αγοράς, το δυναμικό της χαρακτήρα, το πόσο τηλεπικοινωνίες μας έχουν τάσεις ανάπτυξης τότε ε, είναι κάτι που είναι ευρέως γνωστό. Η Ευρώπη καθυστερεί. Έχει μείνει πίσω. Εάν δεν λάβουμε μέτρα γρήγορα να δράσουμε, είναι σαν να ετοιμάζουμε το δρόμο μας για την οικονομική παρακμή. ...όπως είχε υποθεί και πριν από λίγες δεκαετίες... γενικώ για την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχουν ε, κάποιες προτάσεις, λίγες απλές ιδέες... που θα ήθελα να σας αναπτύξω σήμερα για να ομορφύνουμε αυτό το τοπίο. Ένα τοπίο που είναι κατακαιρματισμένο προς στιγμή. <clears throat> Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας στην Ευρώπη ως προς την αγορά του ραδιοφάσματος είναι ένα τερατούργημα Έχουμε 28 διαφορετικές αγορές, η κάθε μια είναι σαν τη χιονάτη με τους 7 νάνους και υπάρχουν 100 προμηθευτές η Ευρώπη. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ανταγωνιστική, αλλά στην πραγματικότητα η κατάσταση αυτή το μόνο που δημιουργεί είναι σύγχυση. Ολιγοπόλια, περιορισμοί Θα ήθελα λοιπόν να κάνω δύο προτάσεις. Προτάσεις για να πάρουμε την κατεύθυνση της προόδου. Να δημιουργηθεί επιτέλους μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Ε, είναι σημαντικό να συζητήσουμε πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση στην κατανομή του φάσματος όλη την Ευρώπη και στο σχετικό χρονοδιάγραμμα ακόμη και αν δεν ανοίξει τελείως η αγορά, είναι σημαντικό να ε, γίνει κοινό ο μηχανισμός και ακόμη και αν δεν γίνει αυτό πλήρω, πρέπει να συντονιστούμε, να συντονίσουμε περισσότερα από όσα γίνονται τώρα. Η κατανομή του φάσματος να ε, γίνει βάση συντονισμού. Είναι σημαντικό αυτό προ την κατεύθυνση της ενιαία αγοράς τηλεπικοινωνιών. Δεύτερη παρατήρηση. Κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό. Γιατί κάποια στιγμή χάσαμε την αίσθηση της πραγματικότητας και αρχίσαμε τις δημοπρασίες για την ε, ε, απόδοση του ραδιοφάσματος. Αυτό πρέπει να πάψει. Οι φορείς τηλεπικοινωνιών θα πρέπει επιτέλους να πάψουν να πληρώνουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασίες, σε πωλήσει ουσιαστικά, ραδιοφάσματος και μετά να δυσκολεύονται να επενδύσουν. Να επενδύσουν και να χτίσουν τα σημαντικά. Το πραγματικό δίκτυο των τηλεπικοινωνιών. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διερευνήσουμε άλλους τρόπους, όπως κάποια κράτη μέλη έχουν κάνει άφε αυτών τους, να έχουμε αιτήσια τέλη για τη χρήση ραδιοφάσματος, ίσως να παραμείνουν οι αγοραπολισίες όσοι είχαν, γιατί είναι τελείως θεμητό κάτι τέτοιο στον εμπορικό τομέα, αλλά με άλλο τρόπο να διοργανωθεί αυτό. Δηλαδή να μην επιβάλλουμε αυτό το απίστευτο κόστος, αυτό το τεράστιο βάρος στις εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Είναι τεράστιο αυτό το βάρος, διότι πραγματικά χρειάζονται τα χρήματα οι αρχές, αλλά θα έχουν ακόμη περισσότερα αν επιτρέψουμε στις εταιρείες τηλεπικοινωνία να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να φτιάχνουν δίκτυα, όχι δίκτυα μάλλον, όχι να αγοράζουν ε, μερίδια ρεδιοφάσματο για να τα αποδώσουν στους πελάτες τους. Και τελευταίο, επιχει... τελευταίο σημείο, ένα επιχείρημα που πολύ συχνά προβάλλεται σε ό,τι αφορά το γιατί έχουμε δυσκολίες να λαμβάνουμε αποφάσεις στον ε, χώρο του φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβαίνει αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες καταστάσεις παγιωμένες σε κάποιες χώρες και είναι δύσκολο να αλλάξουν μέσα στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η πρότασή μου λοιπόν θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα διευθυντικά ταμεία για να καταπραίνουμε την μετάβαση των χωρών αυτών, να διευκολύνουμε τη μετάβασή τους, προς την εναρμονισμένη κατανομή του ραδιοφάσματος προκειμένου να υπάρξει σύγκληση, προκειμένου όλα τα κράτη-μέλη να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση με παρόμοια ταχύτητα προς την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Eh, Ευχαριστούμε πολύ. Αγγίξαμε και πάλι ένα σημείο ζωτική σημασία για την ε, κατεύθυνσή μας προ μια εσωτερική αγορά που να είναι ανταγωνιστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Είδαμε το θέμα από διαφορετικές σκοπιές. Θα ήθελα λοιπόν σε πρώτη φάση να δώσω στους συναδέλφους το λόγο για να δούμε τι θέλουν να σχολιάσουν από την πρόταση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ασχολούμαστε με το τμήμα αυτού του φάσματος, το οποίο εναρμονίστηκε για την χρήση των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών. Εδώ μιλάμε λοιπόν για την πολιτική του ραδιοφάσματος, αλλά όχι γενικά. Για τα θέματα αυτά υπήρξε ούτως ή άλλως ε, συζήτηση και πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για το κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο του ραδιοφάσματος. για τομείς που δεν αφορούν τις ε, τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες συγκεκριμένα, μπορεί να επηρεάζονται από το στόχο της πρόταση αυτή ω προς το φάσμα, αλλά δεν μιλάμε ακριβώ για αυτά. Σε κάποιε από τι αιτιολογικέ σκέψει υπάρχει κάποια σχετική επιμονή και θα επιμείνω και εγώ στην ανάγκη να υπάρξει άνοιγμα και άλλων τμήματων του φάσματος, ιδίως της συχνότητας 700. Και εφόσον βρισκόμαστε σε μια επιτροπή που ασχολείται με τέτοια θέματα, θα πρέπει στο σώμα του κειμένου να φροντίσουμε ο κανονισμός να μην περιλαμβάνει πάρα πολλά ε, στοιχεία για τα γενικά προβλήματα που μπορεί να προκληθούν. Την ε, πολιτιστική ε, πολυμορφία, την τις διαφορετικές ανάγκες, όχι γιατί είναι κανονισμός, μιλάμε για άμεση ισχύ σε διαστολή με μια οδηγία. Και άλλο πράγμα η γνωμοδότηση, άλλο πράγμα η έκθεση. Δεν πρέπει εδώ να φανούμε ασυνεπείς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το περιεχόμενο ενός τέτοιου νομοθετικού οργάνου να πλατιάζει Μην ξεχνάμε λοιπόν τον πρωταρχικό στόχο αυτής της πρότασης νομοθεσίας. Το λέω γιατί κοιτάζω και τον πίνακα περιεχομένων όσα αναφέρονται ως τίτλοι τον broadcast. Θα έλεγα λοιπόν να μην επιμείνετε σε αυτά τα στοιχεία, αλλά να θυμόμαστε πάντοτε τον ακριβή στόχο αυτής της νομοθετικής πρότασης. Εναρμονισμένη χρήση του φάσματος για τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες. Συμφωνώ πάντως με αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κάποια βήματα πρόοδου ως προς τη διάρκεια των δικαιωμάτων στο εναρμονισμένο φάσμα προτείνεται η διάρκεια να μην είναι κατώτερη των 30 ετών. Για τα υπάρχοντα τμήματα του φάσματος που είναι ήδη ενεργονισμένα. Ιδάλλως, διερωτώμεθα τι γίνεται με όσους ε, έχουν δικαίωμα για 30 χρόνια αλλά έχουν καταβάλει το τίμημα για τη μισή διάρκεια. Νομίζω λοιπόν ότι το επιπλέον φάσμα ε, θα μπορούν να το λάβουν χρονικά εφόσον το ξεπληρώσουν κιόλα. Βέβαια, εδώ θα μπορούν οι εθνικοί ρυθμιστέ να κάνουν τι προτάσεις τους. Εγώ, σε συγχέτρια, δεν μπορώ να το προκαθορίσω. Αυτό θα επιληθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλά νομίζω είναι λογικό να υπάρξει παράταση της διορίας σε σχέση με αυτό που αρχικά Νομίζω πάντως ότι το να παραταθεί η διορία είναι κάτι που δεν θα πρέπει να καταλήξει στο να υπάρξει ένα μέσο το οποίο να μην αξιοποιείται. Μιλάμε για την αγορά φάσματος. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα δυναμικότερο χαρακτήρα στην αγορά του φάσματος. Μου φαίνεται και αυτό ενδιαφέρον. Μιλάμε για κίνητρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και όπως είπαν στις παρατηρήσεις τους οι συμμετέχοντες, μέχρι τώρα λείπουν. Φαίνεται εδώ λοιπόν ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών είναι κάτι που ίσως και να ε, γίνει περιττό εφόσον αυτό που επιδιώκουμε είναι περισσότερες σχέσεις συνεργασίας. Εάν κάποιος δεν συμφωνεί μπορεί να πάρει ένα άλλο τόνο του φάσματος. Μια και φτάσαμε ως εδώ, να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Κατρίν. Oui, euh, Μία παρατήρηση σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στον κανονισμό αλλά και στην μέθοδο. Βεβαίω, εγώ ε, λέω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια περίμετρος αναφοράς ε, στον κανονισμό όμως η Κομισιόν δεν δίστασε να βάλει πολλά πράγματα και μάλιστα με προβληματικό τρόπο ε, όσον αφορά ε, την ισχύουσα οικονομική ρύθμιση. Ε, πρέπει να σεβαστούμε βεβαίως μια μεθοδολογία συγκεκριμένη. Ωστόσο θα πρέπει να βάλουμε και μια τάξη στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Αυτή είναι η άποψή μου, την έχω πει άλλωστε και επανειλημμένα, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, όσον αφορά τώρα το φάσμα. Ξεκινήσαμε με τον ορισμό ε, μιας ε, συντονισμένης διαδικασίας ε, των κρατών μελών για πιο εναρμονισμένη διαχείριση του φάσματος. Διαπιστώνω ότι ο κατάλογος που είχε προβλεφθεί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πρέπει να τον δούμε έτσι ώστε να κάνουμε συζήτηση όσον αφορά την οικονομική, το οικονομικό βάρος του υφιστάμενου φάσματος και του μελλοντικού φάσματος. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνένεση, αλλά ε, πρέπει να, πάρουμε και μια, να κάνουμε και μια στρατηγική επιλογή. Ε, το Κοινοβούλιο ασχολείται με το φάσμα ε, κυρίως απέναντι στον δισταγμό του Συμβουλίου, ενώ ξέρουμε, όπως το υπενθύμισε και ο καθηγητής κ. Πογκορέλ, ξέρουμε την οικονομική σημασία του φάσματος. Είναι οικονομικός παράγοντα. Επομένως, ποιο είναι ο βαθμός συντονισμού με το υφιστάμενο πεδίο όσον αφορά και την δευτερογενή αγορά. Ε, ε, τι θα κάνουμε, τι προβλέπετε. Δεύτερον, σε περίπτωση κατά την οποία ε, έχουμε ευθυγραμμισμένο ε, ημερολόγιο ας πούμε απόδοσης φάσματος σε όλες τις χώρες τι θα γίνει με τους βιομηχάνους ε, και νομίζω ότι εδώ αναφέρθηκε στο τελευταίε στις τελευταίες παρατηρήσεις και η Πιλάρ Καστίγιο γιατί στην ουσία θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου αγοράζουν ε, φάσματα σε κάποιες χώρες τις οποίες τα οποία πληρώνουν αργότερα, έτσι είναι η κατάσταση τώρα, θα περάσουμε λέω στην κατάσταση όπου θα πρέπει το φάσμα να πληρώνεται ε, άμεσα. Ε, δηλαδή ακολουθούμε διαφορετική οικονομική οδό και νομίζω ότι δεν έχει ληφθεί αυτή η διαφορά αρκετά υπόψη και όσον αφορά την πρόσβαση και όσον αφορά και την πληρωμή πρέπει να βρούμε κάποια λύση η ετήσια πληρωμή θα μπορούσε να διευρυνθεί. Ε, μπορούμε να σκεφτούμε όμως και κάποια άλλα συστήματα, όχι μόνο την μηνιαία καταβολή. η ε, ενεργοποίηση της αγοράς οπωσδήποτε περνάει από την αποσαφήνιση των ε, δευτερογενών αγορών και επίσης το κόστος ε, που μπορεί να είναι δυσβάσταχτο για τις ε, επιχειρήσεις αντιπροσωπεύει και τον τρόπο ε, με τον οποίο μπορεί κανείς να περάσει σε ένα πιο εναρμονισμένο φάσμα και βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα αντιδράσουν τη στιγμή που θα πρέπει να αγοράσουν το φάσμα και που θα πρέπει να περάσουν και στις ίνες ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Στη Νότια Κορέα έμαθα περνούν ήδη στην επόμενη ταχύτητα. 5G για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων. Φαίνεται πως χρειάζονται τότε συντομότερα διαστήματα ανάμεσα στα κέντρα μετάδοσης, δηλαδή και πιο πολλές αντένες ίσως ε, και λοιπά. Υπάρχει αυτό ως εναλλακτική επιλογή για να επανέλθουμε στο ραδιοφάσμα ή όχι. Άλλες ερωτήσεις σας παρακαλώ, λέει η κυρία Ντελ Καστίγιο. Ο κύριος Κανέλος. Έχω μία διπλή ερώτηση. Μία προς την κατεύθυνση του εκπροσώπου Deutsche Telekom και η άλλη προς τον κύριο Πογκορέλ. Εμείς στην Μπερέκ θα θέλαμε να βάλουμε και business enablers και να δράσουμε ως business enablers δηλαδή στην αγορά και να δώσουμε το φάσμα που χρειάζονται οι operator χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δυναμική της αγοράς ούτε την οικονομική σταθερότητα των operator. Κατανοώ ότι ορισμένοι μεγάλοι operator όπως η δική σας εταιρεία ε, αντιμετώπισαν δυσάρεστες εκπλήξεις σε ορισμένες δημοπρασίες φάσματος, σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, επειδή η Κομισιόν προτείνει τώρα το streamlining του φάσματος υπό ορισμένε προϋποθέσεις, θα ήταν η επιχείρησή σας διατεθειμένη να δαπανίσει εκατομμύρια σε ταυτόχρονες δημοπρασίες σε, το, σε ολόκληρη την Ευρώπη για να περάσει το φάσμα των 700 MHz. Δεύτερη ερώτηση προς τον καθηγητή Πογκορέλ. Κατανοώ καλά ότι αυτό που εννοήσατε ήταν να χαμηλώσει η τιμή πρόσβασης στο φάσμα με αντάλλαγμα καλύτερες υποχρώσεις κάλυψης, για παράδειγμα σε υπαίθριε περιοχέ όπω έκαναν ορισμένε χώρε όπω η Γερμανία και η Σουηδία, θεωρείτε ότι αυτό είναι μια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή για να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στι υποχρεώσει κάλυψη και στην ε, πρόσβαση στο φάσμα. Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα τα μέλη του πάνελ να μπορέσουν να απαντήσουν, λέει η κυρία Ντέλ Καστίγιο. Ευχαριστώ. Να απαντήσω λοιπόν και εγώ στα γερμανικά. Τουλάχιστον ένα μέρο των ερωτήσεων μου τέθηκε στα γερμανικά και πρώτα για την περαιτέρω εξέλιξη Έχουμε ένα οδικό χάρτη της διεθνούς διεθνών προδιαγραφών. Αυτό το 4G, το LTE δηλαδή, το οποίο υπόκειται στον οδικό αυτό χάρτη. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι περί το 2016 θα μπούμε στην επόμενη φάση, AT Advanced, και αυτή η επόμενη φάση θα χρησιμοποιεί και περισσότερο φάσμα καθώς επίσης και με εφαρμογή άλλων μέτρων θα είναι σε θέση να επιτύχει πολύ υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης. Και το 5G θα έλθει 2-3 χρόνια αργότερα. Αυτά που βλέπουμε σήμερα λοιπόν είναι και έχουν και την έννοια των τεστ. Δεν είναι εφαρμογή του 5G ακόμα. Άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Για το LTE Advanced δεν είναι νέο, δεν νέα προδιαγραφή, νέο στάνταρτ. Είναι ένα σύνολο μέτρων που εφαρμόζονται, για παράδειγμα περισσότερη τεχνική κεραιών και άλλα, spectrum aggregation που σημαίνει παίρνω τμήματα φασμάτων για παράδειγμα 800, 1800, 900 και 2000 και εικονικά τα συνδέω ώστε να επιτύχω υψηλότερη ταχύτητα και ευρύτερο φάσμα. Ρωτήσατε επίσης πώς θα καλυφθεί η μελλοντική έξτρα ζήτηση. Έχουμε στην επόμενη ΔΕΑΣΕ 15 ζήτημα της ημερήσιας διάταξης για να βρούμε νέο, να εντοπίσουμε νέο φάσμα βίαση και οι σχετικές ομάδες εργασίας, οι εθνικές δηλαδή, εργάζονται από αυτού και στην ΔΕΑΣΕ 15 θα μπορέσουμε για την IMT να ξεύρουμε νέο φάσμα. Σε ό,τι αφορά το ραδιοφάσμα, είπα και πριν ότι θεωρούμε ότι η Ευρώπη θα εναρμονιστεί με τις παγκόσμιες κατανομές θα συμμετάσχει δηλαδή και η απόφαση που λήφθηκε στην WAC 12 θα ισχύσει και αυτή που μπαίνει και αυτή μέσα στο ευρυφάσμα. Δεν βλέπω όμως την μεγάλη σύγκρουση με το ραδιόφωνο που συχνά ακούμε, διότι την λύση της σύγκρουσης αυτής την βλέπω να περνά μέσα από την timeline. Όποιος δηλαδή στη βάση της σημερινής ζήτησης, αλλά και με τις μελέτες που είναι γνωστές. Η ζήτηση λέει ότι το 2016 με 2018 δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τη ζήτηση με τα φάσματα που έχουμε σήμερα. Βέβαια το ραδιόφωνο χρειάζεται και κάποιο χρόνο για να μπορέσει να αντιδράσει στις διάφορες χώρες μέλη για να μπορέσει να εφαρμόσει και πιο σύγχρονες προδιαγραφές και για να καθαρίσει το φάσμα θα μπορέσουμε νομίζω να συμφωνήσουμε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο ώστε όλες αυτές οι δίθεν απειλούμενες συγκρούσεις τελικά μάλλον δεν θα επισυμβούν. Μια ερώτηση κάνατε ακόμα για τις πανευρωπαϊκές δημοπρασίες αν θα θέλαμε δηλαδή να συμμετάσχουμε ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Δεν είμαστε όμως παρόντες σε όλες τις αγορές και οι άλλοι operator το ίδιο. Δεν έχουμε λοιπόν ίχνος σε όλη την Ευρώπη των 28. Επομένως εναρμονισμένες συνθήκες είναι σημαντικό να μην μπορούν οι διάφορες χώρες μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές συνθήκες ή να αφήνουν κάποιους ε, συμβούλους να τους τις επιβάλλουν ενώ οι ίδιες οι χώρες δεν τα κατανοούν τόσο καλά τα πράγματα αυτά για να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά θα έχουμε ένα set of rules, εναρμονισμένους κανονισμούς δηλαδή. και που θα ελέγχονται και από την Ευρώπη με εναρμονισμένο τρόπο. Αν γίνει αυτό, τότε δεν χρειαζόμαστε ταυτόχρονε ε, δημοπρασίες σε όλες τις χώρες μέλη. Αρκεί να είναι εναρμονισμένοι οι κανόνες, οι συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Η Νίκολα και μετά ο καθηγητής Μπογκορέλ. Α, εσεί πρώτο, πρώτο κύριε καθηγητά, εσείς, ναι. Ναι, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να διευκρινίσω ε, πάλι ορισμένα πράγματα. Αυτό που σκέπτομαι πέρα από την ισορροπία αυτή μεταξύ κάλυψης και τελών για το φάσμα. Ακούμε συχνά ότι ορισμένες χωρισμένοι μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να συγκλίνουν τα σχέδια συχνοτήτων τους, ιδίως νέες χώρες μέλη έχουν δυσκολίες για να συγκλίνουν τα σχέδια συχνοτήτων τους με τα σχέδια συχνοτήτων άλλων χωρών, παλαιότερων χωρών μελών. Η πρόταση εν προκειμένου είναι να βοηθήσουμε όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης να προχωρήσουν προς τα μπρος στην ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ταχύτητα για να γίνει αυτό να χρησιμοποιηθούν τα διαθωτικά ταμεία για να τους επιτρέψουν να αναδιασκευάσουν τον σχεδιασμό συχνοτήτων τους. Αυτό νομίζω θα είναι μια πραγματικά ριζοσπαστική προσέγγιση για να τους επιτρέψει να φτιάξουν την σίλικον ε, αυτή αγορά στην Ευρώπη. Η Νίκολα. Σας ευχαριστώ. Για να απαντήσω πρώτα στην ίδια την Πιλάρ. Κατανοούμε ότι οι κανόνες που προτείνονται εδώ είναι για το ροδιοφάσμα. που έχει εναρμονιστεί για την ασύρματη επικοινωνία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιεί το ίδιο από άλλους χρήστες προηγουμένως. Η διαδικασία εγκατάλειψης του φάσματος, καθαρισμού του φάσματος, πρέπει να υπακούει σε κάποιες ρυθμιστικές αρχές, με την έννοια των principles, που έχουν μπει και στο πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Αυτή τη διευκρίνηση προτείνουμε εμείς. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό του εναρμονισμένου φάσματος θα πρέπει να μπει και αυτό στο πακέτο. Τι σημαίνει εναρμονισμένο φάσμα. Δεν διευρύνουμε δηλαδή το πεδίο εφαρμογής, αλλά διευκρινίζουμε τους όρους. Ακούσαμε πριν λίγο, και είναι σωστό βέβαια, ότι η media distribution γίνεται όλο και περισσότερο επιγραμμικά. Όμως, σύμφωνα με τα νούμερα που διαθέτουμε, και είναι ενδιαφέρον αυτό, η τηλεόραση για 93% εξακολουθεί να είναι live. Υπάρχει ένα 5% μαγνητοσκοπημένων ε, εκπομπών και 2% μόνο είναι επιγραμμικά, που μεγαλώνει μεν, αλλά μεγαλώνει σιγά σιγά. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, ούτε θεωρούμε ότι θα μεγαλώσει ξαφνικά στο μέλλον. Και είναι σαφές ότι η παρακολούθηση ζωντανής τηλεόρασης στο διαδίκτυο, αν πάνε όλοι στο ευρύ φάσμα, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν θα είναι δυνατόν πλέον να παρακολουθήσουν όλοι ζωντανά τηλεόραση επιγραμμικά. Γι' αυτό λέμε ότι η ψηφιακή χερσαία πλατφόρμα εξακολουθεί να είναι πιο αποτελεσματική και για το επόμενο θέμα, το οποίο επίσης αναφέρθηκε, η σύγκριση στη χρήση στην ε, καλωδιακή τηλεόραση όπου έχετε το τηλεοπτικό σήμα που έρχεται μαζί με την επιγραμμική πρόσβαση, πάλι εκεί εμείς ζητούμε αποτελεσματικό, συνδυασμό του broadcasting και της ε, broadband για τη ζωντανή την παρακολούθηση ζωντανής τηλεόρασης ο broadcast mode εξακολουθεί να είναι πιο αποτελεσματικός από το ευρύ φάσμα και νομίζω ότι περισσότερο θα συμφωνήσουν είπες ακόμη ότι θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο φάσμα στο μέλλον. Εμείς δεν είμαστε επεπισμένες, θεωρούμε ότι ακόμα πρέπει να αποδειχθεί αυτό, η ανάγκη δηλαδή περισσότερου ευρέως φάσματος. Μίλησε η κυρία και για την ε, συνέργεια και πρέπει όντως να αποδειχθεί η ανάγκη ότι χρειάζεται δηλαδή παραπάνω ε, ευρύ φάσμα. Νομίζω πρέπει να περάσουμε στο επόμενο πανέλ. Και στο τέλος θα έχουμε άφθονο χρόνο. Για να πάρετε το λόγο όσοι θέλετε. Προχωρήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μάρκους πρώτος είχε πάρει το λόγο προηγουμένως, διευθυντής της WIC. Μετά Φιτόρη, διευθυντής της ΕΚΤΑ και κύριος Μπελτρά της ΜΠΕΟΚ. Κύριε Μάρκους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καστίγιο. Ε, πάντα είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι εδώ. Ε, σήμερα θα σας παρουσιάσω μία σύνοψη ε, της ε, τελευταίας από τρεις ε, μελέτες με το θέμα αυτό. Πολλά από τα σημεία τα οποία θα αναφέρω θα τα βρείτε ήδη στις, ε, ε, στις εκθέσεις ε, αυτές. Επίσης να πω ότι η κυρία Γκάρμποβιτς είναι κοντά μου. Ναι, εδώ λίγο πιο πίσω. Υπάρχει το νέο άρθρο 4α, το οποίο αφορά την δημιουργία συμμαχιών ε, περιαγωγής ε, και που θα προετοιμάσουν τις χώρες ε, για την μετάβαση στο επόμενο στάδιο και βεβαίως με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν νέες τιμές ελευθερία από τους περιορισμούς των τιμών και καλύτερο ανταγωνισμό. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις επίσης θα οδηγήσουν υποτίθεται σε μείωση των τιμών κυρίω περιεγωγής, ε, κυρίως όσον αφορά την μη χρέωση των ε, εισερχομένων φωνητικών κλήσεων. Uh, ε, το, η πρόθεση είναι οι, σταθε, οι κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα να είναι η ίδια με την εγχώρια χρήση των, της κινητής τηλεφωνίας. Ε, η μείωση των τιμών των ε, κλίσεων περιαγωγής ε, που θα πλησιάσουν τις τιμές της εγχώριας κλίσης βεβαίως δημιουργεί κάποια ζητήματα. Ε, είναι, ε, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι αυτές οι roaming alliances του άρθρου 4α θα δώσουν αυτήν την ε, επιδιωκόμενη ελευθερία. Είναι γεγονός ότι τα συμφέροντα των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών δεν είναι ίδια και επομένως αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ενδεχομένως θα υπάρξει ελευθερία από ελέγχους και θα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιοι operators οι οποίοι δεν θα χρειάζονται χρειάζεται πλέον ε, να ε, ε, δώσουν και τις δομικές λύσεις στήριξης του που είναι υποχρεωμένοι να δίνουν μέχρι τώρα. Η πρόταση της Κομισιόν λοιπόν στην ουσία δυναμητίζει μέχρι ένα βαθμό την καλή χρήση της αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προβλέπουμε ότι αυτές οι alliances δεν θα λειτουργήσουν πάρα πολύ καλά. Τώρα, ε, είναι σημαντικό να ε, πούμε ότι η, η μείωση των τιμών λιανικής και χονδρικής ε, είναι πάντα συνδεδεμένες. Για να βρεθεί κάποια τιμή κατά την έννοια της, της μηδενικής χρέωσης για τις ερχόμενες κλήσεις θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα λεγόμενα termination rates, κόστος ολοκλήρωσης κλήσης δηλαδή. Η, προτινόμενη όμως οδηγία, δεν το... κανονισμό συγγνώμη, δεν το κάνει. Ε, ε, ε, υπάρχει μία χονδρική τιμή η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την λιανική τιμή από το ένα δίκτυο στο άλλο. Όσον αφορά τις ε, εισερχόμενες ε, κλήσεις, εδώ δεν ε, προτείνεται πληρωμή για αυτή καθε αυτή την κλήση, αλλά προτείνεται κόστος για την ολοκλήρωση της κλήσης. η διαφορά όσον αφορά την ολοκλήρωση της, το, το κόστος ολοκλήρωσης κλήσης ε, είναι ότι αυτό το κόστος ε, είναι κρίσιμης ε, σημασίας. Η Κομισιόν εδώ και χρόνια προσπαθεί να μικρύνει την απόσταση ανάμεσα στο κόστος της εισερχόμενης κλήσης και το κόστος ολοκλήρωσης κλήσης καθώς επίσης και το, της εξερχόμενης κλήσης σε κατάσταση περιαγωγής αλλά εάν ε, δεν γίνει με σωστό τρόπο, τότε για κάθε κλίση ε, θα υπάρχει κόστος το οποίο θα πληρώνει ο operator της τάξης των τριών ε, cents. Το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κόστος το οποίο προκύπτει σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και οι εθνικές κλήσεις υπό τον νέο κανονισμό θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται σε ξεχωριστούς κανονισμούς από ό,τι, ε, από περιαγωγή. Δηλαδή στην ουσία θα έχουμε τέσσερις ε, κανονισμούς, ε, τέσσερα νομοθετήματα τα οποία θα αφορούν την κινητή τηλεφωνία. Στην προκείμενη περίπτωση των, του κόστους περιαγωγής διεθνών κλίσεων πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αντί να βελτιώσει την αγορά. Αυτό που θεωρούμε εμείς είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε με, με ολοκληρωμένο τρόπο λάβει υπόψη της Κομισιόν στις προτάσεις της και το ε, τέλος ε, της ολοκλήρωσης ε, κλήσης. Και βεβαίως να πω εδώ ότι συμφωνούμε απολύτως με την ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνει η εισηγήτρια για την ολοκλήρωση της κλήσης. Ε, μας ε, απασχόλησε το σύνολο της ε, πρότασης όσον αφορά τις επιπτώσεις. Η κυρία Ντεκαστήγιο ανέφερε ότι η απλούστευση είναι σημαντική. Ένα από τα καλά του παρόντο συστήματος είναι ότι είναι αρκετά ιεραρχημένο. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα κανονισμό για, πραγματικό κανονισμό για την ε, συνδεδεμένη ε, Ήπειρο είναι να ξεκαθαριστεί ακόμα περισσότερο και να συνδυαστούν οι υπάρχουσες οδηγίες και οι μοναδικές οδηγίες μεταξύ τους γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε σε μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχουμε τώρα. Είναι σημαντικό βέβαια να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία τα οποία έχει η πρόταση της Κομισιόν, να μην πετάξουμε το μωρό μαζί με το, με το νερό που του κάναμε μπάνιο. Ε, και βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχημένη εφαρμογή ε, των προτινόμενων μέτρων ε, και να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με καλή ανάλυση. Η έκθεση δικαστήριο πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Φιτόρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μια πολύ ευχάριστη στιγμή η πρόσκλησή σας για να σας παρουσιάσω τις απόψεις του κλάδου μας. Να πω ότι στηρίζουμε το συνολικό στόχο ως έκτα για να ε, μειωθούν οι πιέσεις προς τους χρήστες, ε, οι περιορισμοί και να υπάρξει θετική ε, θετικό κλίμα για τους διασυνοριακούς καταναλωτές. συμφωνούμε με την ιδέα ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση μιας ε, ενιαίας αγοράς, αλλά με συνθήκες ανταγωνισμού, ώστε να μπορούν οι προμηθευτές που έχουν τεράστιο αποτύπωμα ήδη στην Ευρώπη να ανταγωνιστούν μεταξύ τους αποτελεσματικά. Ωστόσο, είναι σημαντικό ο κλάδος να έχει και νομική βεβαιότητα και να υπάρχει προβλεψιμότητα ε, σε σχέση με τους ε, εφαρμοστέους κανόνες αλλά και με το τι επενδύσεις χρειάζονται για να μπορεί κανείς να συμμορφούται με τους κανόνες. Προς στιγμήν υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, προτάσεις για λύσεις επιτάπητος, νομικός δεσμευτική ε, πρόταση στον ε, κανονισμό περιαγωγή 3 οι οποίες επιβάλλουν τη συμμόρφωση των εταιριών έως το 2014. Γιατί οι διαφορετικές αυτές εναλλακτικές οδηγούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Διότι αν οι φορείς, οι προμηθευτές, μειώσουν τα τέλη της περιαγωγής με ένα ευθυγραμμισμένο σύστημα, ε, ένα ενιαίο σύστημα αντί για το decoupling ή αν η περιαγωγή καταργηθεί ε, βάση νομοθεσία έω το 2016, τότε το decoupling και η σχετική υποχρέωση θα καταστεί καινή νοήματος. Το decoupling, η αποσύνδεση, δημιουργήθηκε στην αρχή για να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες ανταγωνισμού και οι δυνάμεις της αγοράς να μειώσουν και να περιορίσουν τα τέλη περιεγωγής. Αλλά αν τα ίδια τέλη ε, εξαλειφθούν με άλλες ε, μεθόδους, το να επενδύει κανείς πια στην αποσύνδεση δεν θα έχει νόημα, θα είναι περιττό και θα είναι μια ε, ανόητη επιπλοκή. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ο κλάδος ζητά και εκλυπαρεί τους πολιτικούς ηθήνοντες να κάνει λογικές επενδύσεις, να υποχρεώσει σε λογικές επενδύσεις μέσω των νομοθετικών ε, μέτρων. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη και έχει ήδη αναφερθεί είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν καταργήσουμε τα τέλη περιαγωγής βασινόμου, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ούτως ή άλλως θα υπάρχουν ε, τα θα υπάρχει το κόστος της ε, όπως το τέλος της παύσης. Αυτό κάπως θα πρέπει να το αντισταθμίσει ο κλάδος. Ίσως να είναι αρνητικό το αποτέλεσμα από την σκοπιά των καταναλωτών αλλά εάν οι καταναλωτέ που δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίε περιαγωγή πρέπει να πληρώσουν τη ζημιά, δηλαδή να αντιεπιδοτήσουν, ε, να αντισταθμίσουν το κόστος που επιβάλλουν οι υπόλοιποι καταναλωτές που ταξιδεύουν διασυνοριακά, αυτό δεν θα είναι πολύ δίκαιο και δεν είναι καθόλου διαφανές ούτε και φιλικό προς τον ε, τελικό χρήστη, τον καταναλωτή. Τελική μου παρατήρηση είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε το εξή. Εάν τα τέλη περιαγωγής καταργηθούν βάσει νόμου, όπως προτείνει η συγκήτρια, τότε θα πρέπει αυτό να ακολουθηθεί από κανόνα δίκαιης χρήσης. Λίγο πολύ στις γραμμές της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή Ήτρε που προσκαλεί την οργάνωσή μας Ευρωπαίων Καταναλωτών για να, σημα... για να συζητήσει το σημαντικό αυτό θέμα. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών. Καταναλωτών. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα άνω των 40 οργανώσεων σε πάνω από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Συμφωνούμε με την κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει μια κίνηση για την μείωση των εθνικών φραγμών για την περιαγωγή που ζητούμε εμείς εδώ και πολλά χρόνια να ζητηθούν να μειωθούν τα τέλη. Η περιαγωγή όσο οι καταναλωτές γίνονται πιο κινητικοί γίνεται και πιο σημαντική. Θέλω να επενθυμίσω το ψήφισμα 2593 του 2013 για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης και μέσα εκεί λέει ότι μέτρα τα οποία θα ολοκληρώσουν την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να οδηγήσουν στο κλείσιμο των κενών ε, μέχρι το 2015 για, με κατάργηση των τελών περιαγωγής. Ζητούμε από τους συνομοθέτες με την ευκαιρία αυτή που ανοίγεται σήμερα να λάβουν τα μέτρα αυτά που θα επιτύχουν ακριβώς αυτό. Η πρόταση της Κομισιόν λοιπόν έχει τον στόχο Ε, έχει θετικό αποτέλεσμα από, του, από την άποψη ε, των καταναλωτών. Όμως ο μηχανισμός προτείνει το 4α μας ανησυχεί για δύο λόγους. Πρώτον, ο προτινόμενος μηχανισμός για συλλογικές συμφωνίες θα έχει σημαντική επίπτωση στον ανταγωνισμό και επομένως στην ε, ποιότητα και ποσότητα της επιλογής που θα έχουν οι καταναλωτές. Για ορισμένους operator με ορισμένο μέγεθος, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να αποτελέσει μόνο κίνητρο χωρίς κανένα αντικίνητρο. Το δεύτερο το γεγονός ότι προβλέπονται και γεωγραφικά κριτήρια μπορεί να οδηγήσουν σε μια Ευρώπη δυο ταχυτήτων όπου ορισμένοι θα υποφελούνται και άλλοι όχι. Εξαρτάται δε αυτό από τη χώρα τους και από το ποιος είναι ο operator. Εν τέλει η ανάλυση που κάνουμε εμείς είναι ότι ο προτινόμενος μηχανισμός είναι υπερβολικά περίπλοκος χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και ενδέχεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στους καταναλωτές και δυσπιστία απέναντι στους μηχανισμούς περιαγωγής. Εάν η αγορά δεν επιτύχει λοιπόν να ρυθμίσει το θέμα, θεωρούμε ότι οι συνομοθέτες θα πρέπει να ακούσουν ε, αυτά που λέει το Κοινοβούλιο και να καταργήσουν τα τέλη περιαγωγή μέχρι το 2015. Η δε συζήτηση πρέπει να στραφεί γύρω από το πώ θα το επιτύχουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι οι οροφέ της περιαγωγή του 2012 δεν ήταν αρκετές. Η πρόταση της Κομισιόν μειώνει το κόστος για την λήψη τηλεφωνημάτων, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ιδίω τα beta caps έχουν μείνει πολύ πίσω και δεν έχουν μειωθεί αρκετά. Επίσης με την ευκαιρία αυτή θέλω, όπως είπε ο κύριος Μάρκους προηγουμένως, να πω και εγώ ότι με τον στόχο δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς, οι διασυνοριακές υπηρεσίες, δηλαδή το έξτρα κόστος, πρέπει να καταργηθεί. Ενιαία αγορά χωρίς φραγμούς για τον καταναλωτή. Το να σε μέλος της οικογένειάς σου λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα, πρέπει να είναι το ίδιο φτηνό όσο να πάρει τηλέφωνο του γειτονά σου. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι είναι ανεξήγητα ακριβέ αυτέ οι υπηρεσίε και πολύ μακριά από το να κλείσουν το κενό που τις χωρίζει με τις εγχώριες υπηρεσίες. Γι' αυτό ζητούμε να επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ε, υπηρεσίε αυτέ χωρί. να καθίσουν να σκεφτούν αν ο συνομιλητής του βρίσκεται σε άλλη χώρα μέλο Μόνο τότε θα έχουμε φτάσει σε πραγματική ενιαία αγορά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς κύριε Μπελτρά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ένα γύρο ερωτήσεων-απαντήσεων. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην ε, Επιτροπή, στην Επιτροπή Περιφερειών Έχουμε και εκπρόσωπο της ΕΟ και όχι, όχι δεν έχουμε, δεν μπόρεσα να έρθει και μετά και στο κοινό. Θα ήθελα να κάνω τις εξής διευκρινήσεις όσον αφορά τη δικιά μου πρόταση για την περιαγωγή. Εν πρώτης, Το ζήτημα είναι ότι ξεκινάμε από μία ε, κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει η περιαγωγή είναι vintage πλέον. Είναι vintage product πλέον. Είναι επεπαλαιωμένο. Εδώ και 7 χρόνια ε, παλεύουμε με κανονισμούς ε, για την ε, περιαγωγή. Και το αποτέλεσμα μιλήσανε, πέσανε λίγο οι τιμές και τα λοιπά. Έχουμε roaming 1, roaming 2, roaming 3 και ε, μπορεί να συνεχίσουμε με νομοθετήματα τα οποία θα αφορούν την περιαγωγή, θα αυξάνεται ο αριθμός των νομοθετημάτων για να μειώνεται σιγά σιγά και λίγο η τιμή. Εμείς θέλουμε να εξαφανιστεί το, η περιαγωγή, το roaming ε, βεβαίως γιατί θα είναι οικονομικό συμφέρον των ε, πολιτών που ταξιδεύουν, αλλά θα είναι επίσης, θα έχει επίσης και συμβολική έννοια. Θα αρθεί, θα εξαφανιστεί ένα σύνορο, ένα όριο το οποίο, το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μόλις φύγεις, βγεις από τα σύνορα της χώρας σου, η χρήση του τηλεφώνου ή το, της ταμπλέτας ή ε, η, ε, η χρήση δεδομένων, η, η αποστολή μηνύματος ή δεδομένων γίνεται εξαιρετικά περίπλοκο πράγμα. Ε, δηλαδή γίνεται πιο περίπλοκη η ζωή μας με το που περνάμε τα σύνορα. Τότε τι έννοια έχει που είμαστε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέμε ότι οι διασυνδέσεις θα πρέπει να είναι ε, απλές. Εδώ δεν είναι ούτε απλές ούτε φτηνές. Επομένως, εάν το κόστος αυτό μειωθεί, εάν ληφθούν αποφάσεις τέτοιες που να ε, ε, μειώσουν το κόστος της περιαγωγής, βεβαίως αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Τη μέρα που ένας πολίτης της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας ή της Γερμανίας ή της Πολωνίας ή οπουδήποτε αλλού από την Ευρωπαϊκή Ένωση σηκώνει το τηλέφωνο και τηλεφωνεί στο σπίτι του ή παίρνει την ταμπλέτα του και ε, τον υπολογιστή του και χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, τότε αλλάζει η αντίληψη για την Ενωμένη Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι το απτό. Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένη ότι θα αποτελέσει ένα απτό σημάδι, ένα απτό μήνυμα που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όλα τα μέρη του κόσμου ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη πραγματικά δημιουργούμε μια εσωτερική αγορά και αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Όχι μόνο για τους χρήστες, έναν γενικό οικονομικό αντίκτυπο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι απαιτείται πολιτική απόφαση. Μία συγκεκριμένη στιγμή δηλαδή να πούμε ότι τελείωσε, δεν υπάρχει πια αυτό το σύστημα. Περνάμε σε άλλο κεφάλαιο. Μετά από 7 χρόνια απανοτούς κανονισμούς νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ε, ε βεβαίως θα πρέπει να είναι ε, σαφές το θέμα της ασφάλειας δικαίου. Εάν ε, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τώρα το θέμα αυτό, δεν θα το καλύψουμε ποτέ. Είναι πολύ συγκεκριμένο και άπτεται άμεσα ενός συστήματος συγκεκριμένου που ε, λειτουργεί με βάση την νομική ασφάλεια. Λοιπόν, λέμε ας πούμε ότι σταματάει η επιπλέον χρέωση των, ε, της περιαγωγής ή των εισερχόμενων ε, κλήσεων. Εδώ και ένα χρόνο το, το λέμε αυτό. Ε, και θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν λέω να διατηρηθεί η νομική ασφάλεια. Εγώ δεν είπα ούτε το 2014 ούτε το 2015. Εγώ είπα το 2016 γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε ε, όλους όσους προσπαθούν να αναπτύξουν ε, τέτοιες ε, σωστές προσφορές. Οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, οι operators κτλ. μου, λένε γιατί να επενδύσουμε τώρα στο decoupling εάν πρόκειται μετά να αλλάξουμε θέση. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε αλλάξει το decoupling ε, νωρίτερα. Εάν δεν λειτουργήσει τουλάχιστον το 2016 το νέο σύστημα ε, roaming. Κανείς δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι αυτό το σύστημα θα λειτουργήσει. Ενδεχομένως θα πρέπει να περιμένουμε και το 2017 και μετά το 2017 να πούμε «Α, πρέπει να το αλλάξουμε». Νομίζω πάντως ότι με την ημερομηνία που επιλέξαμε το 2016 αφήνουμε αρκετό χρόνο στους εμπλεκόμενους φορείς ε, να προχωρήσουν και στις απαραίτητες ε, προσαρμογές και μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και να μην υπάρχουν πλέον καθόλου επιπλέον κόστη περιαγωγής ή θα κρατήσουμε ένα σύστημα διαχωρισμού. Θα το δούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μου φαίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο είναι να καθορίσουμε μια τελική ημερομηνία στην οποία θα εξαφανιστούν αυτά τα τέλη περιαγωγής. Τώρα, σε σχέση με άλλα κόστη del 2015 se haya hecho eh, κόστος χονδρική. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του ορίου, του ενότητα του ορίου, του πλαφών έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε κατά κάποιο τρόπο τις ανάγκες ε, του κλάδου ε, και να δούμε πού μπορεί να βρούμε μια, ένα σημείο ε, ανάμεσα στην χονδρική και στη λιανική. Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μερικά σύντομα σχόλια για τα θέματα που μας παρουσιάσατε και ιδίως για όσα είπατε εσείς μόλις τώρα. Το είπε και ο εκπρόσωπος τον, ε, του Συλλόγου των Καταναλωτών για τα θέματα περιαγωγής. Η περιαγωγή δεν έχει κανένα νόημα. Σε άλλες ανταγωνιστικές οικονομίες με αγορές ακόμη πιο ολοκληρωμένες όπως των ΗΠΑ, πιο ενοποιημένες μάλλον όπως των ΗΠΑ, η αγορά είναι πολύ πιο ζωντανή. Η πρόεδρος έκανε λόγο για την έννοια μιας εσωτερικής αγοράς με τεράστιο οικονομικό δυναμικό, όμως η περιαγωγή είναι και πολιτικό ζήτημα. Γιατί, γιατί εγκρίναμε το πακέτο περιαγωγή 3 και ο Ευρωπαίος πολίτης Προσπαθεί να καταλάβει τι κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Ίσως είναι ένα μήνυμα μόνο, αλλά είναι σημαντικό να ακουστεί. Ε, είναι πολιτικό το θέμα. Και ε, είναι σαν να επιδιώκουμε με την τρόπο αυτό και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εάν λοιπόν πραγματικά θέλουμε εσωτερική ενιαία αγορά για τις τηλεπικοινωνίες, η περιαγωγή δεν έχει πια κανένα νόημα. αλλά θα συμφωνήσω με την Πιλάρντε Καστίγιο. Πρέπει να φροντίσουμε και την νομική βεβαιότητα. Να έχουν οι επενδυτές την ασφάλεια ότι μπορούν να επενδύσουν. Ε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε δια όλα. Ο κύριος Μάρκους είπε ότι χρειάζονται ξεκάθαρα δεδομένα. Δεν είναι βέβαιο το τι θα συμβεί αν πάει κανεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα όταν ταξιδεύει. Οπότε το πρώτο που τον απασχολεί είναι να αποσυνδέσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να αναζητήσει ένα hotspot για το ίντερνετ, για το wifi. Δεν βρίσκω όμω ότι είναι η καλύτερη φόρμουλα αυτή. Σε ευχαριστώ, Σαλβαντόρ. Άλλε ερωτήσεις από του συναδέλφου αλλιώ να δώσω το λόγο στου ομιλητές και να περάσουμε στο τελικό τμήμα της συνεδρίασης, της ακρόασης, χωρίς ε, πλέον καθυστερήσει. Okay, uh, Ίσως να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση πρώτα. Τι θα γίνει με την αυξημένη χρήση όταν ταξιδεύουν οι πολίτες και πώς αυτό έχει συσχετιστεί με την αλλαγή στις τιμέ. Για τα τηλεφωνήματα δεν αρκεί. Για τα δεδομένα ίσω, Με τη μελέτη ενδεικτή που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδαμε μετά την υλοποίηση του κανονισμού από το 2012 και από όσα έγραψε ένας ε, εξέχων οικονομολόγος, ο κ. Μπέρντινγκ, ότι ήταν μείον 2,4 το ποσοστό αντί για μείον 2,7 ε, που είχα υπολογίσει εγώ. Δεν έπεσα και πολύ έξω και σίγουρα είναι καλύτερο από το ποσοστό για τα δεδομένα που μάλλον ε, από αυτό που θα γινόταν αν δεν είχε εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Και για τα δεδομένα ε, εντοπίστηκε ότι ευτυχώς έχουν μειωθεί τιμές. Η ελαστικότητα φτάνει το μείον 1%. Εάν λοιπόν τα τέλη περιεχογή μειωθούν για τα δεδομένα, έχουν μειωθεί ούτω ή άλλω από το 2011 χρονιά για την οποία μελετήθηκαν τα δεδομένα. Τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα. Αλλά ευτυχώ τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα για τα δεδομένα από ό,τι είναι για τα ε, φωνητικά. Άλλο κανεί. Άλλη παρέμβαση γι' αυτό. Εσείς. που μα δίνετε την ευκαιρία θα μιλήσω και εγώ ισπανικά και ήθελα να πω το εξή. αναφερόμενο σε αυτά που εξηγήσατε κύριε Τελικαστήγιο και πρώτα συμφωνώ όταν λέτε ότι η κατάργηση της περιαγωγής έχει και συμβολικό χαρακτήρα αλλά οι διαμεθοριακές κλήσεις, ε, οι διεθνείς κλήσεις δηλαδή, είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Είτε πρόκειται για Γάλλους, είτε πρόκειται για Ισπανούς, το ίδιο πράγμα είναι. Οι διεθνείς κλήσεις είναι σημαντικές για την ενιαία αγορά. Εμείς ασφαλώς είμαστε υπέρ της ασφάλειας δικαίου. Το επιχείρημα είναι ισχυρό και σίγουρα το αναζητεί ο κλάδος. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε λόγο αυτό το decoupling να είναι δήθεν ασυμβίβαστο με την περιαγωγή. Και μάλιστα θεωρούμε ότι θα κινηθεί στο ίδιο επίπεδο όπως για την εγχώρια αγορά. Ναι, κύριε Δικαστήριο, γι' αυτό που είπατε τώρα στο τέλος θα εξαρτηθεί από το πώς θα γίνει το decoupling, από την αποδοτικότητά του θα εξαρτηθεί αν θα λειτουργήσει ή όχι. Αλλά αυτό το ξέρουμε ακόμη. Πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα πάει. Για να μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό, να το αξιολογήσουμε δηλαδή, ε, χρειάζεται να περάσει κάποιο χρόνο. Αυτό που λέω εγώ για ασφάλεια δικαίου είναι κάτι διαφορετικό. Ασφάλεια δικαίου σημαίνει ότι χρειάζεται μια εύλογη προθεσμία για τις προσαρμογές για τα διάφορα έργα και επίσης για να δοκιμαστούν αυτά. Αλλά για την αποσύνδεση ακόμη δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα αποδώσει και η διεθνή κρίση είναι άλλη ιστορία πάλι, διότι εκεί η αγορά δεν είναι ρυθμισμένη. Μιλούμε για άλλο πράγμα επομένως. Άρα, όπως είπα και πριν, για να είμαι ειλικρινή, οι, οι, οι οικονομικές πτυχές είναι σημαντικές. Σημαντικό είναι να μειωθεί το κόστο ώστε να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες. Όπως είπα όμω και η συμβολική αξία είναι τόσο σημαντική που αναμένω πολλά θετικά από αυτό. Βέβαια, εάν ε, γίνει αυτό θα είναι πολιτική απόφαση διότι το business as usual θα σήμαινε απλά ότι αφήνουμε να περάσουν οι ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες και ότι εξακολουθούμε να φορτώνουμε στους πολίτες περί το κόστος. Τώρα η Κομισιόν και μετά η Επιτροπή των Περιφερειών. Έχουμε μέχρι τις 6.30 ακόμη. Και είμαι βεβαία ότι και η Περιφέρεια και, ε, ε, συγνώμη, με και η Κομισιόν και η Επιτροπή των Περιφερειών δεν θα εξαντλήσουν το χρονικό περιθώριο ώστε να μπορέσουν να λάβουν το λόγο πάλι και οι άλλοι. Η Κομισιόν, λοιπόν, πρώτα έχει το λόγο, παρακαλώ. Εισηγήτρια, σκιώδεις εισηγητές, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε. Μας προσκαλέσατε απόψε. Δεν ευχαριστώ για την ακρόαση αυτή όπως συνήθως γίνεται από αυρότητα ή ευγένεια. Αυτά είναι πράγματα που λέγονται συνέχεια και είναι τετριμένα. Όχι, το εννοούμε πραγματικά εγώ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν μια πολύ χρήσιμη μέρα διότι κρατήσαμε πλήθος σημειώσεων, σωρία σημειώσεων και νομίζω ότι πραγματικά μάθαμε πολλά. Μάθαμε πολλά μετά από τη σημερινή συζήτηση αλλά και τη χθεσινή ε, ακρόαση που διοργανώθηκε. Βεβαίω ε, και από ευγένεια σα ευχαριστώ γιατί ευγενικοί άνθρωποι είμαστε, αλλά είναι και ειλικρινεί οι ευχαριστίε μου. Όταν η αντιπρόεδρο Κρού ε, πρότεινε το πακέτο αυτό για τι τηλεπικοινωνίε, πιστεύω ότι ε, πίστευε στην δημοκρατική διαδικασία και είπε ότι η δημοκρατική αυτή διαδικασία θα βελτιώσει την πρότασή μας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ε, υποβάλαμε μια αρχική πρόταση και συνεισφέρουμε μαζί με όλους τους ε, ενδιαφερομένους σε μια διαδικασία που είμαι βέβαιος ότι εσείς ως συνομοθέτες θα την κάνετε να ξεχωρίσει, ε, να θα φροντίσετε να βελτιωθεί η αρχική μας πρόταση και θα κάνετε καλή δουλειά για αυτό το σκοπό. Αυτό το αποδεικνύει και η σημερινή ακρόαση και βρισκόμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την τόσο κοπιαστική πορεία των τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ίσως όχι τόσο κοπιαστική, πάντως είπε ότι είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη και ότι θα μετατρέψει με όποιο τρόπο μπορεί την ευρωπαϊκή οικονομία σε ψηφιακή οικονομία και ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να ξεφύγουμε από το οικονομικό τέλμα και να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Ένα άλλο πολύ σημαντικό βήμα είναι οι δύο επαγγελματικότατε εκθέσει των δύο εισηγητών του Κοινοβουλίου, ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ. Ε, οι επιτροπές, οι εισηγητές των επιτροπών αυτών μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές τους και όλους τους συνεργάτες τους συνεισέφεραν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Ειλικρινώς αυτό που έγινε χθε, αλλά κυρίως σήμερα, πραγματικά άλλαξε την θεώρησή μας για το πακέτο Connected Continent. ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων που ήταν αμφιλεγόμενο. Κάποιοι είχαν αμφισβητήσει τη χρησιμότητά της. Κάποιες φορές ε, κορόιδευαν και παρουσίαζαν ε, σαν καρικατούρα την πρόταση αυτή. Άκουσα βέβαια διαφορετικές ε, μεταφράσεις από τα ακουστικά μου και διαφορετικές γλώσσες, αλλά όλοι είπαν τον όρο σύγκληση. Σύγκληση σε σχέση με αυτό το πακέτο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσω πολύ και τον πρόεδρο του Μπέρεκ, ε, η οποία συνεισφέρει τα μάλα στην όλη αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εσάς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, ο χρόνο δεν είναι πάντοτε με το πλευρό μα. Ε, θα χρειαστούν προανελημμένε διαβουλεύσει και στην πρωτοδοτικού σα φορέα, όμω πραγματικά σα ευχαριστώ. Και η συμβολή των ενδιαφερομένων ε, φορέων σε αυτό το στόχο ήταν πολύ σημαντική, αλλά κυρίως το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικότατο ρόλο, επισημένοντας πολύ ε, εύστοχα ζητήματα τα οποία πρέπει να μελετηθούν. Ήταν επικοδομητική λοιπόν η στάση σας. Πάντως, στη φάση αυτή δεν έχω καμία ε, εξουσία ή αρμοδιότητα να προτείνω συμβιβαστικές λύσεις ή να συμβιβάσω διαφορετικές απόψεις, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι ακριβής στα σχόλια που θα κάνω σε σχέση με όσα ακούστηκαν. Έχω δικαίωμα να πω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλη αυτή τη διαδικασία θα φανεί ανοιχτόμυαλη, διαλλακτική και ε, θα φροντίσει να ακουστούν όλες οι απόψεις προκειμένου να επιλέξει την, τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό για να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Αυτό το είπε και αντιπρόεδρος Κρούς και το επαναλαμβάνω. Τώρα για να σταθώ στα διάφορα σημεία που σχολιάστηκα, που συζητήθηκαν σήμερα βλέπουμε ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας γενικότερης συμφωνίας, σύγκλησης απόψεων για το πώς πρέπει να διοργανώσουμε τις υπηρεσίες του διαδικτύου και το φάσμα. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο αποτέλεσμα. Ήδη είδαμε ε, στις εκθέσεις των εισηγητών ε, ΙΜΚΟ και ΙΤΡΕ ενδιαφέρουσες ιδέες, άλλες επίσης ενδιαφέρουσες ιδέες πρέκυψαν χθε και σήμερα. Από όλα αυτά έχουμε μια πολύ καλή, πλούσια βάση για να προχωρήσουμε. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτό. Για την ενιαία ε, αδειοδότηση. Να πω το εξής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία συναισθηματική προσκόλληση σε κάποια λύση ή εις βάρος κάποιες άλλες. Ο στόχο είναι να υπάρχει μια εταιρεία που να προσφέρει υπηρεσίες χωρίς να, να καταβάλει υπερβολικά ψηλούς να μην εκβιάζεται καμία εταιρεία από κράτη-μέλη που λένε ότι θα σας άρω την άδεια, θα σα την αναστείλω εάν ε, δεν συμμορφωθείτε με τους κανόνες μου, δεν, εφόσον υπάρξει κάποια σοβαρή παραβίαση, βεβαίω αυτό μπορεί να γίνει, αλλά όχι ως πολιτική δράση. Θα πρέπει μια εταιρεία, εφόσον λαμβάνει αδειοδότηση, να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της παντού στην Ευρώπη. Η εισηγήτρια είπε ότι οι ιδέες για την απλούσταση της διαδικασίας και η Μπέρεκ νομίζω συμφωνεί με αυτό, ε, είναι οι καλύτερες και θα το εξετάσουμε με πνεύμα, όπως σας είπα, διαλλακτικό, ανοιχτό και ε, προκειμένου να μπορέσουν οι εταιρείε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παντού. Με όσο το δυνατόν πιο ταχύς ρυθμούς και αποτελεσματικά. Αυτό που θα προκύψει από την όλη συζήτηση θέλουμε να ε, το εξετάσουμε με, μεγάλη, με τη δέουσα προσοχή. Ε, υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν καλωσορίζουμε τη συζήτηση που έγινε. Επίσης πρέπει να επαναλάβω, ξανά και ξανά ίσως θα έπρεπε να το πω, και το έχω ξανακάνει, αλλά αξίζει να το επαναλάβει κανείς, πουθενά δεν λέγεται στην πρόταση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευνοεί τη μία λύση εις βάρος κάποιων άλλων λύσεων. Όχι, αυτό που προτείνεται είναι μια πρόταση αρχή, μια αρχή που, που προτείνουμε. Δηλαδή ότι οι ρυθμιστές θα πρέπει να επιλέξουν την αναλογικότερη ε, λύση δεδομένων των ρυθμιστικών συνθήκων στο κάθε κατός Εάν κάποιο, κάποιο μέσο είναι αναλογικότερο από κάποιο άλλο, το ψηφιακό δηλαδή σε σχέση με το υλικό, θα μπορούσε να επιλεγεί το ένα ή το άλλο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κράτου μέλου. Μια άλλη ψευδέστηση σε σχέση με την πρόταση είναι ότι επιβάλλεται μια ενιαία για όλους λύση. Δεν αληθεύει αυτό σε σχέση με την πρόταση. Λέει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινό μοντέλο για τα εικονικά προϊόντα. Ακούσατε ε, τις απόψεις ε, του επιχειρηματικού κόσμου απόψεις που είναι πολύ σημαντικές, αλλά υπάρχουν και άλλες φωνές. Ε, η δημόσια δίκηση, το νέφος, όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Να σας παραπέμψω στη μελέτη που εκπονήθηκε πριν από δύο χρόνια για για το κόστος της μη Ευρώπης. Η σύσταση που ακούστηκε είναι ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλα αυτά τα προϊόντα. Ε, εκπλήσουμε λοιπόν κάποιος, ε, εκπλήσουμε κάπως που κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή έκανε τέτοιου είδους πρόταση. Σημειώνουμε και καταγράφουμε ότι η Μπέρεκ θέλει να το επεξεργαστούμε το θέμα αυτό. Αλλά στο ε, πνεύμα συνεργασίας που μας διέπει θα το κάνουμε. Όμως η κριτική για το SSF θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν από πάρα πολύ καιρό. Δεν έγιναν όλα αυτά που θέλαμε, εντάξει, αλλά ας το επιτρέψουμε. Ας το επιτρέψουμε, διότι αν τώρα έχει ε, ξεχαστεί και το αφήσουμε κατά μέρο, θα χάσουμε άλλα δύο χρόνια. Υπάρχει όμω και ενδιάμεση οδό. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του Connected Continent, τη ε, ε, υπήρου στο διαδίκτυο. Δεν είναι ιδανικό βεβαίω το σενάριο που προκύπτει, δεν είναι το σενάριο τη πρόταση, αλλά είναι ένα σενάριο που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά θα συνεργαστούμε, θα συνεργαστούμε και μαζί σας και με το Συμβούλιο και οι ιδέες που ακούστηκαν σήμερα και σαφείς ήταν και ε, καταλάβαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε δεν είναι αναγκαστικά αυτός που αναφέρεται ως προς την διακυβέρνηση, governance, πρέπει να πω ότι σκοπός μας ήταν να ενισχύσουμε την ΠΕΡΕΚ. Να είναι ισχυρή και ανεξάρτητη. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη δήλωση του Προέδρου της Μπέρεκ και στην επόμενη Ολομέλεια θα κοιτάξουμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια μόνιμη θέση Προέδρου στην Μπέρεκ ευχαρίστως να ακούσουμε τις συζητήσεις που θα γίνουν στην ΠΕΡΕΚ και ελπίζω ότι εδώ και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο θα τα λάβουν αυτά υπόψη. Για την περιαγωγή. Καλωσορίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας να εργαστούμε και στα θέματα του roaming. Αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό ζητά και κατά πρώτον το Κοινοβούλιο με το ψήφισμα που ενέκρινε πρόσφατα, αλλά και η Επίτροπος Κρούς, αυτά είπαν προσφάτως. Το, ε, ως προς την περιαγωγή, δεν ε, είναι λογικό να πρέπει κανείς συνεχώς να αποσυνδέει τις ταμπλέτες του, τα κινητά του τι θα κάνουμε με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα στο μέλλον, θα τα κλείνουμε στα ε, σύνορα. Η περιαγωγή είναι ένα στοιχείο του παρελθόντος, Αυτό είναι σαφές, Προέκυψε και μέσα από τη συζήτησή μας. Όμως υπάρχει ένα σημείο ε, επί του οποίου διαφωνούμε ίσω με κάποιους από τους ομιλητές. Το τέλος του roaming δεν θα πρέπει να είναι ε, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη ρύθμιση. Αυτό θα ήταν παράδοξο. Ο μόνος τρόπος να τελειώνουμε τον περιαγωγή είναι να μην αυξήσουμε τη ρύθμιση. Διότι τότε θα εκτροχιαστούμε. Πρέπει τη λύση να τη βρει ο ίδιος ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών μπορούμε να το εξετάσουμε, μπορούμε να συλλογιστούμε, μπορούμε να βρούμε μια καταληκτική, μια προθεσμία μάλλον, αλλά εάν θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος στο, στην περιαγωγή, θα πρέπει να μην επιβάλλουμε περαιτέρω ρυθμιστική πίεση για, τις διεθνείς, για τα διεθνή για τις διεθνείς κλήσεις, νομίζω ότι πρέπει η αγορά όντως να είναι απελευθερωμένη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως, πώς θα αλλάξει η αρχή αυτή μέσω της πρότασής μας. Η πρόταση κάνει, δίνει ιδέες για μέτρα διαφάνειας και αυτά θα αποτελέσουν μέρος του κανονισμού. Ε, ένας καταναλωτής που ξέρει τι να κάνει, θα χρησιμοποιήσει φωνητικές ε, επιλογές, θα χρησιμοποιήσει κάποια πακέτα ε, προσφορών. Στα περισσότερα κατημέλη όμως το 60% των πληθυσμών πληρώνει μειωμένες τιμές για τηλεφωνήματα εντός Ευρώπης. Ε, από την ε, Πορτογαλία Λισαβόνα στο Βίλνιο, στη Λιθουανία, ε, το λεπτό κοστίζει 1,2 ευρώ. Το λεπτό κόστος. Η τιμή είναι 1,2 ευρώ, ενώ το κόστος είναι 3 λεπτά. Εδώ Βλέπουμε λοιπόν τα μέτρα αυτά να μην ε, βασίζονται στην πραγματική, να μην έχουν στόχο να αλλάξουν την τιμή. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνει κάποιες προτάσεις σχετικά η Μπέρεκ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, uh, Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφερειών. Βεβαίως ε, θα βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε σε αυτά ε, αλλά και στο τέλος ε, θα μπορέσουμε παρόλες τις διαφορές να κάνουμε μια καλή πρόταση αλλά για την περιαγωγή ένα πράγμα να δούμε αυτή την λύση που θα προέρχεται από τον κλάδο όχι επειδή δεν πρέπει να γίνει έτσι όχι επειδή ο κλάδος δεν θα πρέπει να εγκύψει περισσότερο στα διάφορα, στις πτυχές του θέματος, αλλά δεν μπορείτε όμως να πείτε στους ψηφοφόρους και στους πολίτες, ακούστε, περιμένετε, περιμένετε. Ναι, ομαλή διαδικασία, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Διότι οι απαιτήσει της χονδρικής μπαίνουν στην πρότασή μου, γι' αυτό το λόγο τις βάζω. Χρειάζεται να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ένα ξεκάθαρο σήμα ότι κάποια μέρα θα αρχίσουν τα πράγματα αυτά να γίνονται. Εφτά χρόνια κανονισμού περιαγωγής δεν θα γίνει δεχτό από τους Ευρωπαίους πολίτες, πολίτες και το κατανοώ. μπορούμε να δώσουμε χρόνο στον κλάδο να τα κάνει όλα αυτά, αλλά το 2016 χρειάζεται να έχουμε ασφάλεια δικαίου και αναμένουμε από την Κομισιόν να ηγηθεί της προσπάθειας ώστε το σχήμα που θα δώσουμε να είναι καθαρό. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, Επιτροπή Περιφερειών. Εσείς, αλλά πέστε το όνομά σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς κυρία εισηγήτρια. Λέγομαι Φρανκ Τσίμερμαν. Είμαι εισηγητή στην Επιτροπή Περιφερειών για το πακέτο τηλεπικοινωνιών και για την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τη δυνατότητα εδώ να σας ακούσω και να μεταφέρω τις απόψεις αυτές όσο γίνεται περισσότερο στη δική μας συζήτηση. Χαίρομαι όμως επίσης για τη διαβεβαίωση της Κομισιόν ότι οι ιδέες που κατατίθενται εδώ θα ληφθούν υπόψη και θα συζητηθούν σε ανοιχτή διαδικασία συζητήσεως όπου και η ίδια η Κομισιόν θα είναι ε, διαθέσιμη προς συζήτηση. Έχω ορισμένες ερωτήσεις κυρία Πρόεδρε που ίσως καταστήσουν ε, σαφέστερη και τη δική μας προσέγγιση. Πρώτα θα ήθελα να συμφωνήσω με την εκπρόσωπο της European Broadcasting Union αλλά και άλλα μέλη που έθεσαν την ερώτηση αν όντως είναι σημαντικό, είναι απαραίτητος ο κανονισμός ή μήπως ήταν καλύτερα να βασιστούμε στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και να το αναπτύξουμε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουμε ρεαλιστικά βήματα και για την εναρμόνιση και για την υπέρβαση του κατακαιρματισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, για να είμαστε ρεαλιστές, ίσως λιγότερο να αποδίδει περισσότερο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές ε, στις ε, χώρες μέλη. Δεύτερη ερώτηση από τη δική μας σκοπιά είναι το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων. Μήπως είναι καλύτερα για να ξεπεραστεί αυτός ο κατακαιρματισμός, αν είναι όντως σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ο κανονισμός, το μέσον του κανονισμού δηλαδή, και να επιβληθεί η ευρωπαϊκή ρύθμιση σε ολόκληρο τον τομέα. Ή μήπως είναι καλύτερα αρχικά να εξετάσουμε την πραγματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που αυτό χρησιμοποιείται αποδοτικά, πού μπορούμε να επιτύχουμε κάποια καλύτερη, αποτελεσματικότερη χρήση και να επιβάλλουμε ρύθμιση σε αυτόν τον τομέα, ενώ στους άλλους τομείς να επιτρέψουμε να υπάρξει μία κοινή εξέλιξη. Εάν δηλαδή η VTB2 είναι δυνατόν να επιτρέψει την μη χρήση μέρους του φάσματος από τους operator είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από άλλους. Χωρίς όμως να βάλουμε κανόνες από τώρα για, για τμήματα του φάσματος που τελικά δεν ξέρουμε αν όντως θα χρησιμοποιηθούν. Τρίτο ερώτημα, πάλι για το φάσμα, αν όντως είναι απαραίτητο και αν είναι και σκόπιμο να πάμε από 20χρονη αδειοδότηση σε 30χρονη. Όπου ενώ στη Γερμανία τουλάχιστον αλλά και αλλού διαμορφώνονται τάσεις τώρα μάλλον μείωσης των ε, χρονικών αυτών περιθωρίων. Ώστε να υπάρξουν και κάποιες τάσεις προς καινοτομία που δεν διευκολύνονται όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη χρονική περίοδος ερώτηση. Δεν είναι δυνατό να επιτραπεί τέτοια συντομότερη αδειοδότηση. Άλλο θέμα, ουδετερότητα του δικτύου. Εμείς ανησυχούμε λίγο ότι με το να επιτραπούν συμφωνίες μεταξύ παρόχων περιεχομένου και χρηστών και, και παρόχων ειδικών υπηρεσιών θα υπάρξει εν μέρη κάποιος αποκλεισμός σε βάρος του συνήθους ελεύθερου δικτύου. Ενώ χρειάζεται ξεκάθαροι ορισμοί για το ποια είναι τα δικαιώματα των ελληνικών χρηστών και ότι αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του διαδικτύου. Δεν βλέπω όμως να είναι τέτοιο το πνεύμα του κανονισμού ακόμη και εδώ ε, θα χρειαστεί να γίνει πιο συγκεκριμένη ρύθμιση. Θα ήθελα να παραμείνω σύντομος και να μην θέσω όλα τα θέματα που θα περιλάβουμε σε μια πρώτη γνωμοδότησή μας. Στην Επιτροπή Περιφερειών θα λάβουμε απόφαση, την οποία θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σίγουρα θα θέσουμε και εκεί κάποια θέματα που μας απασχολούν, αν και βεβαίως ο ρόλος μας είναι μοναχά συμβουλευτικός. Ελπίζουμε ωστόσο να ακουστούν οι απόψεις μας και να ληφθούν υπόψη στην διαδικασία διαμόρφωσης των απόψεών σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε την Κομισιόν, ευχαριστούμε την Επιτροπή των Περιφερειών. Έχουμε λίγο χρόνο ε, για το ακροατήριο για σας, εάν θέλετε να πείτε κάτι. Like to react to any comments or Θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια, θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ και παρακαλώ πολύ να μας συστηθείτε, βεβαίως. Φρανσουά Λεμέγκρο. Εργάζομαι για μια εταιρεία που ίσως δεν τη γνωρίζετε, λέγεται Cogents Communication. Είμαστε TO1 uh, Internet Service Provider, δηλαδή εμείς uh, ασχολούμαστε κυρίως με το transit. Δουλεύουμε πολύ με το Μεξικό αλλά και με πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και 31 χώρες της Ευρώπης. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα μεγάλα κομμάτια του ίντερνετ. Ξέρετε ότι το διαδίκτυο είναι δίκτυο δικτύων. και στην ουσία είμαστε το μεγαλύτερο interconnected ε, network στον κόσμο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να το κάνω. Θέλω να πω δύο λόγια λοιπόν, γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουν, θέλουν να καταλάβουν ότι το ε, ίντερνετ είναι σαν καταράκτης. Υπερχείληση και πτώση η μέση χρήση της ικανότητας στο διαδίκτυο είναι περίπου 20%. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, χωρίς καθόλου να αυξήσουμε την ικανότητα, με την παρούσα ικανότητα, ε, να έχουμε επί ε, αύξηση της χρήσης του ε, διαδικτύου. Προηγουμένως έγινε λόγος για Um, because the only area where you have congestions are within. Προηγουμένως έγινε λόγος για συμφόρηση. Ε, ε, Γενικώ η υγεία του ίντερνετ είναι καλή. Όντω υπάρχουν αυτά τα ε, congestion lines που είναι, δημιουργούν πρόβλημα, ε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα ε, της άσκησης των δικαιωμάτων και της πρόσβασης των χρηστών network management um, η διαχείριση του δικτύου ε, ε, αυτή βασίζεται στην παλαιά αρχή ότι δεν υπάρχει αρκετή ικανότητα και ο τρόπος με τον οποίο έχει την πρόσβαση γίνεται δευτερεύον ζήτημα. Όταν υπάρχει στην ουσία αρκετή ροή, τότε δεν υπάρχει συμφόρηση, άρα δεν χρειάζεται και διαχείριση δικτύου. Όσον αφορά το technical setup, το co-level του διαδικτύου, εκεί που ε, λειτουργούμε εμείς, δεν δημιουργεί πρόβλημα και ούτως ή άλλως... Ε, η εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που ε, μέχρι να μάθει κάποιος ε, τις λεπτομέρειες του ενός κύματος έχει φτάσει το επόμενο. Έλεγα λοιπόν ότι η συμφόρηση ε, είναι κάτι ασαφές. Όσο κατεβαίνει κανείς πιο βαθιά στο σύστημα, στην πρόσβαση, ε, στους providers, ε, στις, ε, στα δίκτυα διανομής, σε περιφερειακά δίκτυα διανομής, τότε αρχίζουν οι δυσκολίες. Γιατί εκεί δεν, είναι, δεν υπάρχει δυνατότητα επιτάχυνσης σε αυτό το επίπεδο. Ο λόγος που ζήτησα να πάρω το λόγο να παρέμβω At a certain είναι ο εξής. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο, ε, συγγνώμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να έχουν μηδενική ανοχή για την συμφόρηση. Και εάν μπορεί να λυθεί το ζήτημα με κάποιες μπριζούλες, με κάποιες ε, ε, μικρές παρεμβάσεις, να γίνει. That's, really the only sort of, um, αυτό είναι το μόνο μήνυμα που θέλω να σας περάσω. Δηλαδή ότι δεν είναι ε, με κανένα τρόπο αποδεκτή η συμφόρηση. Και νομίζω και το Μπέρεκ πρέπει να το καταλάβει αυτό. Πρέπει να δει τι γίνεται με τους εθνικούς ε, ρυθμιστές να δει ότι υπάρχει αυτό το ε, cascade effect, δηλαδή αυτή η επιταχυνόμενη, ας πούμε, το επιταχυνόμενο αποτέλεσμα εν είδη καταράκτη. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να υπάρχει συμφόρηση. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Έχουμε έξι λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Σε έξι λεπτά πρέπει να σταματήσουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, από την Επιτροπή Περιφερειών νομίζω. Ε. Λέω και ο Γκάμπερ από το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών στο Βερολίνο και ήμουν και εμπειρογνώμων για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειών για το συγκεκριμένο θέμα. Ήθελα να επισημάνω ε, άλλη μια φορά το πρόβλημα της καινοτομίας Στις Ηνωμένε Πολιτείες η FCC έκανε το EMC φάσμα ελεύθερο αδειοδοτήσεων. Έχουμε φτάσει ήδη στους ρούτερ στα 3 GB με ταχύτητα μετάδοσης. Εδώ μπαίνει ακόμη το θέμα ότι πολλοί πάροχοι και κινητής τηλεφωνίας κάνουν το data upload για να επιτύχουν μεγαλύτερες ε, ικανότητες μετάδοσης. Στο θέμα αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ του ανοιχτού φάσματος και του, δικτύου, του ελεύθερου δικτύου. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε προκαλούνται πάλι τεχνητές εχμές. Γιατί βλέπουμε όταν 20-30 ρούτερ μπαίνουν σε ένα δίκτυο, πέφτει δραματικά η ταχύτητα. Επομένως, το ανοιχτό φάσμα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη όπως το αδειοδοτημένο φάσμα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε εδώ. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας για την συζήτηση. Ε, μας βοηθήσατε πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που ήρθατε σήμερα εδώ. Long